So, liebe Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε, ώστε να μπορέσουμε να αρχίσουμε. Mm-hmm. Ο Πρόεδρος. Σήμερα το πρωί η σειρά έχει ως εξής. Πρώτα έκθεση Βάισκερμπερ. Έκθεση Αρσένη και μετά Ντέβελο. Θα δώσω το λόγο ευθύ αμέσω στην κυρία Άνια Βάισκερμπερ για να κάνει την εισαγωγή στη γνωμοδότησή της. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισηγητές κλπ. Ήδη έχουμε διεξαγάγει ορισμένες συζητήσεις και πριν από τις θερινές διακοπές και χαίρομαι τώρα για την συζήτηση που θα ακολουθήσει. Η οδηγία έχει σχέση με την προσπάθεια αύξησης της απασχόλησης. Δυστυχώς, ακόμη τώρα, το 1 πέμπτο των υποθέσεων που τίθεται υπόψη του Solvit έχει σχέση με αναγνώριση προσόντων και αυτά μέσα σε πλαίσια τέτοιας ανεργίας είναι σημαντικά. Το ίδιο και η αντιμετώπιση της έλλειψης ειδικευμένων εργαζόμενων. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται βελτίωση η πρόταση της Κομισιόν και όπως είπα αναμένω να ακούσω και τις απόψεις των συναδέλφων μου. Η γνωμοδότησή μου αναφέρεται ιδίω σε, σε επαγγέλματα υγείας, διότι αυτά είναι και της αρμοδιότητάς μας. Και το light motif μου είναι πάντα η ασφάλεια των ασθενών διότι η κινητικότητα μεν είναι επιθυμητή, από την άλλη μεριά ο ασθενής οφείλει, ή μάλλον οφείλουμε να προσφέρουμε στον ασθενή επαρκή προστασία και ασφάλεια. Δυστυχώς στο παρελθόν υπήρξαν περιστατικά όπου ασθενείς υπέστησαν βλάβη στην υγεία τους ή μάλιστα απεβίωσαν λόγω του ότι δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν γλωσσικά με τους επαγγελματίες υγείας. Αυτά λοιπόν, εγώ εδώ περιλαμβάνω ορισμένα κριτήρια για τις εξετάσεις γλώσσας που θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Προβλήματα βλέπω επίσης στην πρόταση της Κομισιόν σχετικά με την εξέταση μιας επίσημης γλώσσας και έχω συζητήσει και με τον Σκιώδη Συγητή αλλά και η κυρία Μπρέπολς μου τόνισε ότι υπάρχουν χώρες μέλη όπως το Βέλγιο αλλά και το Λουξεμβούργο που έχουν πλήρωνες επίσημες γλώσσες. Και εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα. Εδώ πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η διατύπωση τη ε, Κομισιόν. Δηλαδή τι ωφελεί ένας Γερμανός γιατρός που έρχεται στο Βέλγιο να δουλέψει και πάει στο Ολλανδόφωνο μέρος του να γνωρίζει τα γαλλικά. Δεν ωφελεί σε τίποτα. Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα βήμα προς τα εμπρός. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιστατικά και οι κύριοι Λίζε και Γκρότε μου έχουν θέσει υπόψη τέτοια περιστατικά. Οι ιατροί που έχουν απολέσει την άδεια εξασκήσεως στην πατρίδα τους ασκούν το επάγγελμα σε άλλες χώρες. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει ένα σύστημα προειδοποίησης όχι μόνο για γιατρούς και νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, αλλά και για εκείνους που περνούν από τα σχετικά ε, συστήματα αναγνώρισης και λαμβάνουν τελικά την αναγνώριση των προσόντων. Καθώς και πρόσωπα τα οποία, των οποίων η δραστηριότητα έχει κάποια επιρροή στην υγεία. Και, αυτοί, και αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να υπάγονται στο σύστημα έγκυρης προειδοποίησης. Σημαντικό ακόμη είναι και οι υποθέσεις απάτης εκδόλου, για παράδειγμα με πλαστά ε, πιστοποιητικά σπουδών και αυτά πρέπει να περνούν στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Τώρα, αυτό το διαβατήριο, το επαγγελματικό διαβατήριο των εισαγωγικών που είναι και στην καρδιά της πρότασης της Κομισιόν και απευθύνομαι και στην κυρία Ροτ Μπέρεντ, μου φαίνεται καλή ιδέα, είναι και σημαντική πρόταση της Κομισιόν. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να τονιστεί ο εθελοντικός χαρακτήρας αυτού του διαβατηρίου και η χώρα προέλευση και η χώρα υποδοχής πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία αναγνώρισης. Η δε τελική αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων θα πρέπει να διεξάγεται από την χώρα υποδοχής. Με ιδιαίτερα κριτικό πνεύμα βλέπω και αναμένω τις απόψεις των συναδέλφων τις πολύ σύντομε προθεσμίες επεξεργασίας των αιτήσεων που προβλέπονται για τις αρχές. Στην πρόταση της Κομισιόν συνδέεται η αναγνώριση αυτή, ή μάλλον η πολύ σύντομη αυτή προθεσμία αναγνώρισης, με ένα πλάσμα αναγνώρισης. Δηλαδή θεωρείται ότι ή λογίζεται ότι. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές βλάβες της υγεία των ασθενών. Γι' αυτό και πήρα το άρθρο 4 Δέλτα και το διέγραψα. Αυτό περιλαμβάνει αυτό το πλάσμα δικαίου. Κατά τα άλλα, η εισηγήτρια της αρμόδιας επιτουσίας επιτροπής, η κυρία Πανγιώ, κινείται προς παρόμοια κατεύθυνση. Θέλει δηλαδή να επιτύχει αναβολή. Άρα εκεί συμφωνούμε. Το ίδιο συμφωνούμε με την κύρια εισηγήτρια. Βρίσκομαι και για την μερική πρόσβαση. Πάλι όμως για λόγους ασφάλειας των ασθενών. Η μερική πρόσβαση, ιδίως για τα επαγγέλματα υγείας, επισύρει πολλά προβλήματα. Ιδίως εκεί όπου είναι αυτόματη αναγνώριση διότι υπάρχουν ελάχιστες προϋποθέσεις για τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία. Μου φαίνεται εμένα η μερική πρόσβαση, ιδίω για τα τομεακά επαγγέλματα υγείας, ότι δεν είναι πολύ σκόπιμη η ρύθμιση δηλαδή της μερικής πρόσβασης. Και γι' αυτό έχω προβλέψει εξαίρεση από τη μερική πρόσβαση. Εδώ πάντως, ίσως αυτό <clears throat> να σας ευνηδιάσει προερχόμενο από βουλευτή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, που το Λαϊκό Κόμμα βέβαια προβάλλει ιδιαίτερα την ανάγκη κινητικότητα, αν υπάρξουν άλλε πλειοψηφίε πάντω στην Επιτροπή περιβάλλοντο, τότε θα είμαι διατεθειμένη να επιτρέψω πάλι την πρόσβαση στον ασθενή. Αλλά όπω είπα, αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απόψει των άλλων πολιτικών ομάδων. Τώρα, για τι ελάχιστε απαιτήσει για την εκπαίδευση αποτελούν την βάση για την αυτόματη αναγνώριση των τομεακών επαγγελμάτων υγείας. Υπάρχουν αυτές οι ελάχιστες απαιτήσει για γιατρούς, κτηνιάτρους και οδοντιάτρους, καθώς επίσης και νοσηλευτές, μέες, ε, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες. Για τους οδοντιάτρους έγινε μεγάλη συζήτηση και στον κλάδο των οδοντιάτρων και νομίζω ότι η μεγάλη πάντως πλειοψηφία των ενώσεων των επαγγελματιών αυτών είπαν ότι εκτός από τα πέντε χρόνια θα πρέπει να συμπληρώνονται και οι 5.000 ώρε, όπω και για του γιατρού. Εγώ το λαμβάνω υπόψη αυτό. Αν και δεν είναι για μένα key point αυτό, δεν είναι σημείο κλειδί. Και γι' αυτό πάλι περιμένω εδώ να δω τι θα πούνε οι συνάδελφοί μου για του φαρμακοποιού, αλλά και για τι νοσηλεύτριε που θα πω μετά, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Η λίστα δραστηριοτήτων των φαρμακοποιών δεν ανταποκρίνεται πλέον στις απαιτήσει τη σημερινή πραγματικότητα και γι' αυτό έχω κάνει ορισμένε επικαιροποιήσει προ το τέλο ό,τι αφορά τη λίστα δραστηριοτήτων. Καθώ επίση και η υποχρεωτική άσκηση των έξι μηνών θα πρέπει, πρακτική άσκηση δηλαδή, θα πρέπει να εντάσσεται στον κύκλο σπουδών. Αυτό είναι σημαντικό για τι σκανδιναβικέ χώρε. Η Κομισιόν έχει προβλέψει μια άκαμπτη ρύθμιση ότι αυτή η πρακτική εξάσκηση δηλαδή μπορεί να γίνει μόνο σε κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουν την ευχαίρεια οι χώρε μέλη να αποφασίσουν πότε θα την βάλουν αυτή τη ρύθμιση, πότε θα την βάλουν αυτή την εξάσκηση. Και έχω και τη ρήτρα των τριών ετών, την περιέλαβα ξανά δηλαδή για τους ε, φαρμακοποιούς, όπως ήταν στο αρχικό κείμενο, η οποία ρήτρα λέει ότι οι χώρες μέλη δεν είναι υποχρεωμένες για δεν υποχρεωμένε να αναγνωρίσουν τα προσόντα φαρμακοποιών για τρία χρόνια για την ίδρυση νέου φαρμακείου. Δηλαδή ένας φαρμακοποιός έχει εργαστεί τουλάχιστον τρία χρόνια σε μια χώρα μέλος. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να περιληφθεί. Επιτρέψτε μου να μιλήσω μόνο για τις νοσηλεύτριες ακόμα, κύριε Πρόεδρε, θέμα που εξακολουθεί και είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο έχω κάνει πολλές συζητήσεις, η πρόταση της Κομισιόν λέει 12 χρόνια γενική σχολική εκπαίδευση για τις νοσηλεύτερες και νοσηλευτές. Στην Ευρώπη υπάρχουν δύο δυνατότητες. Αφενός 12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης συν ανώτερη εκπαίδευση, είτε από την άλλη 10 χρόνια σχολείο και μετά ε, επαγγελματική εκπαίδευση. Για παράδειγμα σε Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Αυστρία ε, υπάρχει αυτή η ειδική εκπαίδευση που είναι αυτή η διτή εκπαίδευση που αποσκοπεί στην διασύνδεση του επαγγέλματος με την εκπαίδευση. Γιατί εκεί μαθαίνουν και πολλά θεωρητικά μαθήματα. Το χαρακτηριστικό είναι αυτή, όπως είπα, η διασύνδεση μεταξύ επαγγελματο και θεωρίας. Παλαιότερα, τον Νοέμβριο του 2011 δηλαδή, σε ψήφισμα του Κοινοβουλίου, ζητήσαμε να συνυπολογίζεται αυτό το έξτρα θεωρίας που μαθαίνουν οι νέοι. Για την ε, διπλή, για την διτή αυτή εκπαίδευση, έχω να πω ότι είναι πολύ επιτυχημένη. Οι χώρες που την εφαρμόζουν έχουν και πολύ περιορισμένη ανεργία νέων. Γι' αυτό και τάσομε υπέρ Βεβαίω και οι κάτω χώρε και η Μάλτα που αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με τα 10 χρόνια, να γράψουμε τουλάχιστον 10 χρόνια. Έτσι ώστε δίνουμε στις χώρες μέλη τη δυνατότητα, εάν θέλουν, και μου είπαν ότι οι Ιταλοί για παράδειγμα ζητούν, έχουν μάλλον πάνω από 10 χρόνια υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση, φτάνουν στα 13 χρόνια μάλιστα εξακολουθώ και, είμαι, και με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η άποψη των συναδελφών μου. Ευχαριστώ κυρία Βάις Κέρμπερ, οι σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Πυρίλο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για τη δουλειά της, που μας δίνει πολλές ευκαιρίες να προβληματιστούμε. και γενικά για όλα τα θέματα που θέτει προς συζήτηση. Θέλω να σταθώ μόνο σε κάποια σημεία που θεωρώ προτεραιότητας σε αυτό το θέμα. Στις ελάχιστες προϋποθέσεις πρόσβασης για τους, τις νοσοκόμες και τις ΜΕΕΣ, στο, συντροπολογία 32 λέτε ότι θα πρέπει να κρατήσετε ε, στα 10 χρόνια την εκπαίδευση, τη γενική εκπαίδευση πριν αρχίσει κανείς τις σπουδέ του ως νοσοκόμα ημέα. Δεν συμφωνώ. Η Κομισιόν το βάζει στα 12 χρόνια. Η αύξηση των 10 χρόνων, χρόνων στα 12 χρόνια δικαιολογείται με την εξέλιξη στον τομέα της ε, ιατρικής και των παριατρικών ε, επαγγελμάτων και ικανοποιεί. Και μην ξεχνάμε ότι στην ιατρική τώρα έχουμε πολύ πιο περίπλοκες ε, θεραπείες και πιο ανεπιγμένες τεχνολογίες. Ε, είναι σίγουρο ότι ε, πρέπει να έχουν καλή εκπαίδευση οι νοσοκόμες και οι ΜΕΣ. Αλλά είναι σημαντικό να κάνουν την εκπαίδευσή τους να φτάσουν σε μια ηλικία πιο προχωρημένη ούτω ώστε να φτάσουν σε αυτό το επάγγελμα με τα λόγου γνώσεω. Αυτό δεν εξαρτάται δηλαδή από το αν θα κάνουν 12 χρόνια ας πούμε, ε, ε, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Ε, και το βασικό είναι να έχουν και καλή επαφή με τον άρρωστο. Επομένως, θα πρέπει αυτά τα επαγγέλματα να σε θέση ούτω ώστε να ασκήσουν σωστά το επάγγελμά τους για να εξασφαλίσουν την υγεία των πολιτών μας. Δεν νομίζω ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα 10 χρόνια. Ή μάλλον τα 10 χρόνια ισχύουν για αυτούς που θέλουν να κάνουν το επάγγελμα στη χώρα τους και τα 12 για αυτούς που θέλουν να, την, να κάνουν το επάγγελμα σε μια ξένη χώρα. Όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δούμε πώς θα εναρμονίσουμε τις περιόδους αν θέλουμε να έχουμε αναγνώριση των προσόντων. Στην ε, Ιταλία, όπως υπενθύμησε και η συγγήτρια, ε, η δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μου 13 χρόνια. Πώς θα εναρμονίσουμε τις προϋποθέσεις. Δεν καταλαβαίνω. Και επίσης δεν καταλαβαίνω τις αντιρρήσεις σας στην ε, πρόταση της Κομισιόν για το σύστημα ίνι. E έγκαιρης προειδοποίησης. Η πρόταση της Κομισιόν σχολιάζεται μόνο στο εκτιμώντας 22. Τίποτα σχετικό δεν αναφέρεται στα άρθρα. Νομίζουμε ότι η αρχή αυτή θα πρέπει να ενισχυθεί με ένα ειδικό άρθρο. Ούτω ώστε να λέμε στις αρμόδιες αρχές όλων των κρατών μελών ποιος επαγγελματίας δημιουργεί πρόβλημα. Πρέπει να καταλάβουμε επίσης τη λογική των ε, τροπολογιών που προτείνει η συγγήτρια ε, σχετικά με τις κατεξιοδότηση πράξη. Ah, um, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την ισορροπημένη γνωμοδότηση. Είναι καλή αφετηρία συζήτησης. Υπάρχουν τρία θέματα, ε, προσόντα, γλώσσα και ε, προειδοποίηση. Αυτά είναι τα θέματα προτεραιότητας. Η βασική ανησυχία είναι η γλώσσα και η έγκαιρη προειδοποίηση. Τα θέματα αυτά εν μέρη τα έχει αντιμετωπίσει. Ε, στον Εμένο Βασίλειο πρόσφατα είχαμε μια υπόθεση που τονίζει τα, τις ανησυχίες ε, με τα θέματα της ε, υγείας ε, για κάποιους επαγγελματίες υγείας από άλλα κράτη-μέλη. Και όταν λέμε γλώσσα, ε, μιλάμε και για, και για τη γλώσσα κυριολεκτικά αλλά και μεταφορικά. Κάτι μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Παραδείγματο χάρη, ε, ότι, το ότι έχω ας πούμε κάτι μετρώει σαν σαν καρφίτσα, α πούμε, ή σαν βελόνα, δεν σημαίνει ότι πραγματικά, στα αγγλικά δηλαδή, δεν σημαίνει ότι πραγματικά είναι καρφωμένη μια καρφίτσα, μια βελόνα στο, στο πόδι. Μπορεί να σημαίνει ότι έχω τσιμπήματα απλώ. Στα αγγλικά. Επίση, ε, για την αθεώρηση τη προτινόμενη οδηγία, συμφωνώ με την Κομισιόν. Τίποτα στην ε, πρόταση δεν παραβιάζει τα δικαιώματα των ε, εργοδοτών να τσεκάρουν τις γλωσσικές ικανότητες ε, στη διαδικασία πρόληψης, πρόσληψης του επαγγελματία υγείας. Και αυτό ε, λέγει ότι θα πρέπει, λεγόταν μάλλον, ε, ότι θα πρέπει να αφορά τους επαγγελματίες που έχουν μόνο άμεση επαφή με τον ασθενή. Αλλά αυτό διαγράφτηκε. Επίσης, αυτό το σημείο ε, είναι λίγο σκοτεινό. Θα κάνω τροπολογίες. Η... Τα γλωσσικά τεστ επίσης θα πρέπει να τσεκάρουν και να διαμορφώνονται με βάση το σύστημα του κάθε κράτους μέλους. Επίσης, αν πρέπει να γίνονται δωρεάν, αυτό βαραίνει το κράτος ε, μέλος ε, που εισάγει πολλούς τέτοιους επαγγελματίες υγείας. Επίσης, το κόστος αυτό θα πρέπει να είναι λογικό, αναλογικό και να μην ε, δημιουργεί διακρίσεις στα διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την προειδοποίηση που προβλέπει η πρόταση. Ε, νομίζω ότι μειώνει τους κινδύνους ε, να γίνεται μια προσπάθεια του επαγγελματία να βρει την καλύτερη θέση σε όλη την Ευρώπη. Ε, επίσης πρέπει να προειδοπούνται οι αρχές των κρατών μελών σε περίπτωση που έχει διαγραφεί κάποιος από τα επαγγελματικά μητρώα. Αυτά θα προτείνω τροπολογίες και γενικά μ' αρέσει η πρόταση έτσι ως έχει. Κυρία Βρεπόλς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης συζητητής των Πρασίνων. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Βάισβέργερ, την εισηγήτρια και τη γνωμοδότησή της, που πιστεύω ότι είναι μια σαφής και λεπτομερής ε, πρόταση. Περιλαμβάνει διάφορα σημεία. Εγώ θα επικεντρωθώ κυρίως σε δύο σημεία που πιστεύω ότι χρειάζονται περισσότερες επεξηγήσεις στο κείμενο. Όλοι λένε ότι έχει μεγάλη σημασία η ποιότητα στον τομέα της υγείας. Και το λέει και η συγκήτρια ότι όντω τα προσόντα αυτά πρέπει να μπορούν να αποδειχτούν στην πράξη. Όσον αφορά εμένα, από τη μια πρέπει να υπάρχει η σωστή κατάρτιση που να είναι και επαρκής και από την άλλη μεριά να φροντίσουμε ότι γνωρίζουν και αρκετά γλώσσες ώστε εκεί που θα μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμά τους να μπορέσουν και να συνονεθούν με τους ασθενείς. Στη σημερινή πρόταση όμως υπάρχει το εξής πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα, η κατάρτιση των γιατρών. Στο άρθρο 24 λέει η Επιτροπή ότι η ελάχιστη κατάρτιση θα πέσει από 6 στα 5 χρόνια. Στην ε, Φλάνδρα αλλά και στη Βαλονία από φέτος την έχουμε μειώσει από 7 στα 6 χρόνια. Το να γίνει 5 χρόνια τώρα, αυτό να ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια μας θα το κλάβουν πολύ αρνητικά. Γιατί ο κόσμος θα φοβηθεί ότι δεν θα υπάρχει αρκετή κατάρτιση, ότι δηλαδή δεν θα μάθουν όσα πρέπει τα άτομα αυτά, δεν θα έχουν την απαραίτητη επαφή με τα νοσοκομεία. Από την άλλη η ειδικότητα επιμικίνεται. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι σε άλλα κράτη-μέλη οι ανησυχίες να είναι διαφορετικές και θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μήπως μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες για το τι ισχύει σε άλλες χώρες, δηλαδή πού η πανεπιστημιακή εκπαίδευση των γιατρών είναι έξι χρόνια. Και επίσης κάτι άλλο πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Έτσι δεν είναι. Για την πρακτική όμως τι ισχύει, ισχύει κάτι διαφορετικό φαντάζομαι. Τότε μπορεί να μην είναι το πανεπιστήμιο που θα είναι αρμόδιο, αλλά για την θεωρητική εκπαίδευση εννοείται ότι θα πρέπει να είναι πανεπιστημιακή. Εξού και η τροπολογία 30. Κάτι άλλο τώρα είναι οι γλωσσικές ε, απαιτήσει στο 53. Εμείς έχουμε ανταλλάξει απόψεις εδώ στην Επιτροπή αυτή Συμφωνώ ότι για την ασφάλεια των ασθενών πρέπει να υπάρχουν γλωσσικές γνώσεις, να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, δηλαδή τα άτομα του ιατρικού προσωπικού. Το καλοκαίρι σε διάφορες εφημερίδες στη Φλάνδρα εμφανίστηκαν διάφορα άρθρα που αναφέρονται σε αυτή την προβληματική. Το συμπέρασμα είναι ότι εφόσον δεν υπάρχουν γλωσσικές γνώσεις, αυτό οδηγεί σε παρεξηγήσεις και άρα και σε λάθη στην διάγνωση. Στις τροπολογίες της 55 και 56 η συγγήτρια ε, το αναφέρει ότι οι γλωσσικές γνώσεις είναι σημαντικές και πρέπει εκ των προτέρων να ελεγχθούν. Αλλά εγώ θα ήθελα να διευκρινίσουμε ποιες γλώσσες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σαφή σε αυτό. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν εγώ ποιες γλώσσες θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς το ιατρικό προσωπικό της ε, περιοχής, εκεί όπου ασκεί το επάγγελμά του, ο ενδιαφερόμενος ε, ποια ξένη γλώσσα πρέπει να ξέρει. Να ξέρετε ότι είναι μια ανησυχία που δεν υπάρχει μόνο σε εμά, αλλά και σε άλλες χώρες μέλη. Επίσης, για την ειδικότητα θέλω να μου πει περισσότερα πράγματα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η επιμήκυνση έχει να κάνει μόνο για το ακαδημαϊκό κομμάτι της ε, κατάρτισης αυτής ή και για την πρακτική. Ευχαριστώ και για άλλη μια φορά ευχαριστώ την εισηγήτρια και τους σκιώδες εισηγητές. Ο Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Βάις Κέρμπερ για την κατά την άποψή μου πολύ ενδιαφέρουσα γνωμοδότησή της. Μίλησε για τους γιατρούς που χάνουν την άδεια ασκήσεως. Υπήρξε και μια πολύ άσχημη υπόθεση όπου ένας Ολλανδός γιατρός αναγκάστηκε να επιστρέψει την άδεια ασκήσεώς του, μπορούσε όμως, μπόρεσε όμως να συνεχίσει να ασκήσει το επάγγελμά του στην Γερμανία, στην εκλογική μου περιφέρεια που είναι και του Προέδρου. Νομίζω ότι δεν είναι καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει ότι η πρακτική άσκηση, τώρα επιλογή άλλο θέμα, θα είναι στο τέλος ε, των σπουδών. Αυτό είναι ζήτημα επικουρικότητας. Τουλάχιστον δεν θα πρέπει να απαγορεύεται στις χώρες μέλη εφόσον το θεωρούν σωστό να σπάνε την ε, περίοδο πρακτικής ασκήσεως μέσα στις σπουδέ σε πολλά κομμάτια. Άλλο σημαντικό για το δική μου χώρα είναι η εκπαίδευση νοσηλευτριών και μεών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για την ε, Γερμανία. Δεν μπορούμε να δεχθούμε την πρόταση της Κομισιόν και γι' αυτό χαίρομαι πολύ που προτείνει η κυρία Βάις Κέρβερ ε, τροπολογίες. Η ίδια η καγκελάριο κυρία Μέρκελ ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα και μεγάλη πλειοψηφία όλων των επαγγελματικών οργανώσεων στη Γερμανία εμένουν να, να, να επιμείνουμε και εμείς με τη σειρά μα στα 10 χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ ότι ε, στην Γερμανία είναι ε, ανεπαρκείς οι νοσηλεύτριες επειδή μπορούν να αρχίσουν την ε, επαγγελματική τους εκπαίδευση μετά από 10 χρόνια μόνο σχολείου. Εγώ έχω ως γιατρός δουλέψει συχνά με νοσηλεύτριες και έχω εξαιρετικά καλή εντύπωση. Παρακαλώ λοιπόν εδώ να γίνει δεκτή η πρόταση της Άνια Βαρές Κέρμπερ για το συγκεκριμένο σημείο η κυρία Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω όλες και όλους εδώ να προσπαθήσουμε να επανέλθουμε σε αυτό που πρέπει να θεσπίσουμε εδώ, δηλαδή ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν θέλω να απηχείται ούτε η βελγική, ούτε η ιταλική, ούτε η γερμανική νομοθεσία σε αυτό που θα κάνουμε εδώ. Μια, εδώ χρειαζόμαστε μια νομοθεσία που να ισχύσει σε όλες τις χώρες μέλη. Διαβάζω την πρόταση της Κομισιόν, διαβάζω την έκθεση της ε, εισηγητρίας και διαρωτώ με η, πρόταση της Επιτροπής είναι σωστή. Έρχομαι σε αυτό το τελευταίο που είπε ο κύριος Λίζε και που για πολλούς είναι σημαντικό θέμα. Το ζήτημα της σχολικής εκπαίδευσης για τις νοσηλεύτριες. Η κυρία Βάις Κέρβερ θίγει το θέμα στην τροπολογία της υπαρθμών 39. Το λέω αυτό για όσους επιθυμούν να την διαβάσουν. Διαπιστώνω, ή μάλλον θέτω πρώτα το ερώτημα όχι μόνο τα 10 ή 13 χρόνια της γενικής σχολικής εκπαίδευσης, δεν θέλουμε μόνο αυτό το θέμα, αλλά θέλουμε νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια να μπορεί να γίνει μόνος, μόνο, μόνο το πρόσωπο εκείνο το οποίο μπορεί να πάει και στο πανεπιστήμιο, δηλαδή έχει το πλήρες απολυτήριο λυκείου, ας πούμε, στα, το αντίστοιχο στα ελληνικά. Αυτό θέλουμε. Εάν όμως δεν, αν δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε και αυτό υποθέτω ότι δεν είναι αυτό που θέλουμε όλοι εμείς εδώ, Θέλουμε δηλαδή να μπορεί και κάποιος ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει αυτά τα το, το απολυτήριο γιατί τότε 12 χρόνια και τότε ερχόμαστε στο κέριο ερώτημα ότι τα σχολικά συστήματα των χωρών μελών δεν είναι εναρμονισμένα. Έχουμε ορισμένες χώρες μέλη οι οποίες έχουν δύο χρόνια υποχρεωτικά νηπιαγωγείο πριν να αρχίσουν το σχολείο. Άλλα παιδιά, ε, σε άλλες χώρες τα παιδιά πηγαίνουν 6 χρονών στο σχολείο και μετά από δωδεκαετή εκπαίδευση στη Γερμανία μπορούν να προχωρήσουν στο πανεπιστήμιο, αλλά έχουν δύο χρόνια ήδη, προσχολική ηλικία δηλαδή, υποχρεωτικά. Έτσι λοιπόν πάνε μετά από 10 χρόνια στο πρώτο απολυτήριο ας πούμε. Επομένω θεωρώ ότι εδώ η πρόταση τη Κομισιόν δεν είναι επαρκή. Έψαξα να βρω ορισμό τη γενική σχολική εκπαίδευση. Δεν μπόρεσα. Αν την έχετε κάπου καταχωνιάσει, παρακαλώ πέστε μου πού τον ορισμό, τον αν τον έχετε καταχωνιάσει. Πέστε μου πού, γιατί τότε δεν έχετε δουλέψει καθαρά. Πώ είναι τα πράγματα στι 27 χώρε μέλη. Φτιάξτε ένα πίνακα τέλο πάντων. Και τότε θα μπορέσω να συνδιαλεχθώ μαζί σα. Αν όμω δεν το κάνετε αυτό, δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση της Κομισιόν. Δεν την υποστηρίζω την πρόταση της Κομισιόν, διότι δεν εξηγεί πώς είναι η κατάσταση. Δεν γνωρίζω πώς είναι η κατάσταση στην Ιταλία. Ο Πυρίλο λέει 13 χρόνια. Μήπως όμως εδώ περιλαμβάνονται και κάποια χρόνια πριν από το έκτο χρόνο ηλικίας. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένα παιδί στην Ιταλία μπορεί να προχωρήσει σε μια εκπαίδευση μετά τα 19 χρόνια της ηλικίας του. Δεν μπορώ να φανταστώ. Βέβαια, εδώ χρειάζεται κάποια περαιτέρω εργασία για την ώρα υποστηρίζω την τροπολογία τη κυρία Βάσκερμπερ και όχι επειδή αυτή απηχεί την κατάσταση στη Γερμανία, αλλά επειδή θέλω διάκριση να γίνει μεταξύ των ανθρώπων που έχουν το δικαίωμα πλέον να προχωρήσουν σε πανεπιστημιακές σπουδέ και άλλου που προτιμούν να εγκαταλείψουν τη σχολική εκπαίδευση πριν να φτάσουν στο σημείο αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε όλου οπωσδήποτε με απολυτήριο λυκείου, δηλαδή και οι πυροσβέστε πρέπει να έχουν απολυτήριο λυκείου. Τώρα, η Κομισιόν προτείνει στο άρθρο 1 και επόμενα την επαγγελματική ταυτότητα. Που εγώ την υποστηρίζω απολύτω. Εγώ δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια που θέλει να την κάνει οικειοθελή και αυτό που είπε ο κ. Λίζε ότι χάνει την άδεια άσκηση επαγγέλματο ο γιατρό στην Ολλανδία αλλά μπορεί να συνεχίσει να την ασκεί στη Γερμανία. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό εάν είχαμε το επαγγελματικό αυτό διαβατηριό ή ταυτότητα. Με τι δικέ μου τροπολογίε 5, 8 κλπ. Δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια. Το ίδιο δεν συμφωνώ με την εισηγήτρια σε θέματα τις ε, τροπολογίες υπαρχών 50, όπου στην αναγνώριση ορισμένων ιατρικών επαγγελμάτων περιλαμβάνει μόνο τις μισές χώρες. Αυτό ακριβώς δεν θέλουμε. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα επαγγέλματα υγείας που ενδεχομένως είναι πιο εξειδικευμένα σε άλλες χώρες να μπορούν να ε, αναγνωριστούν και στις υπόλοιπες. Γι' αυτό θεωρώ ότι η πρόταση της Κομισιόν είναι καλύτερη. Βέβαια θα χρειαστεί να γίνουν ορισμένε τροποποίησει ακόμη. Και παρακαλώ να συνομιλήσουμε και με τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Ενίας Αγοράς που έχουν σίγουρα κάτι να πούνε προκειμένου. Ευχαριστώ. Καλωσορίζω την ομάδα επισκεπτών από το Ροσκίλντε που είναι προσκεκλημένη της κυρίας Βάλντεμος. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έστερ Έστερ Να μην επαναλάβω όσα έχουν ήδη υποθεί. Αφηρημένα εδώ πέρα μιλάμε για τα 12 χρόνια, 10 χρόνια βάση για την ε, εκπαίδευση. Εγώ όμως θέλω να κάνω πιο συγκεκριμένο το θέμα και να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα για να καταλάβετε ότι η, δεν στέκει πρόταση που έχουμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ας πάμε σε ένα νοσοκομείο στην ε, Ολλανδία. Στην Υπεθρό υπάρχει για τα παιδιά με 30 νοσοκόμους, όπου σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής έχουν περάσει από 4-5 χρόνια εκπαίδευση. Δεν έχει να κάνει με την ποιότητα το θέμα, έχει να κάνει με το ότι μερικές φορές πρόκειται για κάποιον που είναι πίσω από ένα γραφείο και ο οποίος υπογραμμίζει και λέει αυτός ε, πρέπει αυτό, άλλος πρέπει το άλλο. Τώρα μιλάμε για 12 χρόνια γενική εκπαίδευση. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι για μένα περισσότερο σημασία έχει το να κάνει καλά κανείς τη δουλειά του. Και ειλικρινά, μερικέ φορέ κάνουν καλύτερα τη δουλειά του αυτοί που έχουν κάνει 10 χρόνια γενική εκπαίδευση, σχολείο δηλαδή, και μετά έχουν εκπαιδευτεί επιτόπου στο νοσοκομείο, γιατί έτσι έχουν πάρει τι πρακτικέ γνώσει που του χρειάζονται. Αυτοί λοιπόν κάνουν πολύ καλύτερα τη δουλειά του από ό,τι άλλοι που έχουν τελειώσει πανεπιστήμια και οι οποίοι τέσσερα χρόνια ήταν με τη μύτη μέσα στα βιβλία, αλλά μετά φτάνουν χωρί να έχουν κάνει καμία πρακτική εκπαίδευση. Αυτό λοιπόν είναι ένα παράδειγμα που σα δίνω εγώ. Α πούμε, έχει μια νοσοκόμα ένα μωρό στο στο κρεβάτι του παιδιού δίπλα υπάρχει κάποιο που είναι καλύτερα ε, πληρωμένος, ο οποίος έχει περάσει από φοβερές ακαδημαϊκές σπουδές, βλέπει ξαφνικά αίμα στο παιδί ή κάτι συμβαίνει. Αν στην πράξη δεν ξέρει τι να κάνει και πώς να αντιμετωπίσει στην πράξη αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τελικά αυτός ο μεγάλος ακαδημαϊκός πρέπει να έχει περάσει από την πρακτική. Περί αυτού πρόκειται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κοιτάξει τι γίνεται στα νοσοκομεία, στην Ιταλία, αλλού. Πηγαίνετε στα νοσοκομεία και τότε να βγάλετε συμπεράσματα όσον αφορά την κατάρτιση των νοσοκόμων. Αν δεν αλλάξει αυτό, για μένα είναι για τα σκουπίδια. Θέλω ένα καλό σύστημα βέβαια για την κατάρτιση των ε, νοσοκόμων και μια καλή πρόταση. Γι' αυτό επαναλαμβάνω πάει στα σκουπίδια κατά τη γνώμη μου. Η πρόταση αν παραμείνω έχει και δεν αλλάξει. Παρακαλώ σύντομα κυρία Χίπνερ γιατί αλλιώ δεν προλαβαίνουμε, είναι απόλυτα σίγουρο. Και μετά πρώτοι και άλλοι συνάδελφοι. Κρίνω όμω τώρα τον κατάλογο των απολυτών, εντάξει. Κυρία Χίπνερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που πολλοί από τους συναδέλφους συμφωνούν με αυτά που είπαμε εμείς οι Πολωνοί. Το βασικό πρόβλημα στην Πολωνία είναι το θέμα της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των Πολωνέζων νοσοκόμων από άλλα κράτη-μέλη που έλαβαν το δίπλωμά τους πριν ενταχθεί η Πολωνία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με βάση το άρθρο 23 αυτό θα πρέπει να γίνει, με βάση τα προσόντα που έχουν αποκτηθεί. Εδώ όμως, ε, τότε όμως είχαμε ένα διαφορετικό σύστημα. Είχαμε 8 χρόνια ε, σχολικής εκπαίδευσης και μετά 5 χρόνια στη σχολή νοσοκόμων. Αυτές οι γυναίκες είχαν φοβερή πρακτική εξάσκηση, είχαν πάρα πολλές πρακτικές γνώσεις, ήξεραν πραγματικά να φροντίζουν έναν ασθενή, από τα μωρά μέχρι τους ε, γέρους. Δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε αυτές τις νοσοκόμες επειδή έμαθαν, ας πούμε, το, τη δουλειά τους κάτω από ένα διαφορετικό σύστημα. Επίσης το 33.2 θέλω να ανακληθεί. Το άρθρο 30, το 33.3 όμως πρέπει να διατηρηθεί, γιατί μιλάει για την αναγνώριση των ε, διπλωμάτων των Πολωνέζων νοσοκόμων ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διπλώματα που απέκτησαν πριν ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχει αλλάξει βέβαια το σύστημά μας. Έχουμε 10 χρόνια γενικής σχολικής εκπαίδευσης, συν 3 χρόνια πρακτική εξάσκηση. Ούτε αυτό το αναγνωρίζει η Κομισιόν όμως. Γι' αυτό ο εξυγχρονισμός του συστήματος ε, ε, σημαίνει και πιο αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σημαίνει επίσης ότι και οι βασικές ελευθερίες θα είναι πιο αποτελεσματικές, θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά, θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά η εσωτερική αγορά, μόνο όμως εφόσον αναγνωρίζουμε τα προσόντα ανθρώπου που τα απέκτησαν σε ένα άλλο σύστημα. Δεν μπορούμε να τους τιμωρήσουμε επειδή συμμετείχαν σε ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι προτινόμενες αλλαγές νομίζω ότι βρίσκονται στο ύψο των προσδοκιών των πολιτών που περιμένουν ίση μεταχείριση για του εργαζόμενου. Μια στιγμή παρακαλώ και κάτι άλλο. Οι επιπλέον απαιτήσει που ζητάμε από τις Πολωνέζες νοσοκόμους δεν έχουν κανένα, καμία βάση. Θα πρέπει να τι αντιμετωπίζουμε ισότιμα. Και αυτέ οι γυναίκε έχουν αποκτήσει τα ίδια προσόντα. Επίση, με βάση το δικό μα πολωνικό δίκαιο, οι νοσοκόμε αυτέ έχουν το, την υποχρέωση μονίμως να ανανεώνουν τις γνώσεις τους, να ενημερώνονται. Είναι υποχρεωμένες δια νόμου. Ο κύριος Πρόντι. Ε, πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Ιταλική απόφαση δεν ελήφθη στη θεωρία έτσι επειδή μας κάπνισε, αλλά γιατί διαπιστώσαμε κάποια πράγματα. συνολικά το, τα υγειονομικά επαγγέλματα γίνονται όλο και πιο περίπλοκα. Ακόμα και οι νοσοκόμοι λοιπόν θα πρέπει να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές. Χθε ψηφίσαμε τον ορίζοντα 2020. προβλέποντας ριζικές αλλαγές στις θεραπείες, τις ιατρικές είναι αναγκαίο και οι νοσοκόμοι και οι νοσοκόμοι, σε περιπτώσει, να αυξήσουν το περιεχόμενο των γνώσεών τους. Και των θεωρητικών γνώσεων, όχι μόνο των πρακτικών, και των θεωρητικών γνώσεων. Αυτό θέλω να υπενθυμίσω. Ότι, θέλω να πω ότι ο τομέας της υγείας γίνεται όλο και πιο τεχνικός και περίπλοκος. Και ακόμα και οι νοσοκόμοι και ΜΕΣ πρέπει να έχουν μια πιο βαθιά εκπαίδευση και πιο θεωρητική αλλάζει η υγεία. Και επιπλέον, όλο και περισσότερο αποκτούν ε, μεγαλύτερες ευθύνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχει μια δυναμική. Και εγώ πιστεύω ότι είναι λογικό και συνετό και σόφρο να μιλήσουμε για 12 χρόνια. Ίσως και η Ιταλία πρέπει να περάσει τα 13 χρόνια που επιβάλλει τώρα στα 12. Ήδη σήμερα τα συστήματα υγεία, γενικά ο, ο τρόπο που λειτουργεί η υγεία είναι πολύ περίπλοκο. Θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκο στο μέλλον. Ευχαριστώ την συγκεκριά μα, λέει ο κύριο Ζέμπερ, για την εξαιρετική τη εργασία. Συμφωνώ με άλλου συναδέλφου που επέκριναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ιδιαίτερα, λόγω ιδιαίτερα τυπολατρικής πρότασης. Αυτό που έχει σημασία είναι η πράξη, η πρακτική και γνωρίζουμε όλοι ότι χώρες όπως η Γερμανία αλλά και η, Αυστρία, και η Αυστρία έχουν πολύ υψηλές προδιαγραφές, πολύ υψηλά στάνταρτ ε, υπηρεσιών υγείας. Και εκεί βρίσκεται η υπηρεσία που προσφέρεται στον άνθρωπο, στην ασθενή, πραγματικά στο επίκεντρο. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ να έχουμε πανεπιστημιακούς που έχουν αποκτήσει τις γνώσεις τους τα, ε, μελετώντας τα τραπέζια των πανεπιστημίων. Έχουμε ωστόσο καθήκον να βρούμε μια λύση. Αυτό αναμένουν οι πολίτες μας. Η αναγνώριση των, ε, αμοιβή αναγνώριση των κανόνων είναι απαραίτητη για να μπορέσει να λειτουργήσει η ενή αγορά. Και λαμβάνουμε διαρκώς πολλές ε, αναφορές επειδή ακριβώς δεν λειτουργεί το σύστημα αμοιβαία αναγνώρισης. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια ρεαλιστική προσέγγιση όπου να λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη της πρακτικής. Έχουμε κάνει παρόμοια πράγματα και ε, για παράδειγμα για τους ε, βιοτέχνες ή άλλους που ε, ασκούν επαγγέλματα χειρονακτικά αλλά με ειδίκευση. Έχουμε λοιπόν την, μπροστά μας την ανάγκη να κάνουμε μια εναρμόνιση. Το να επιβάλλουμε τώρα πανεπιστημιακό επίπεδο δεν είναι δυνατόν για όλους και οικονομικά αλλά και διότι δεν πρόκειται να προσφέρει καμία βελτίωση στον ασθενή. Διότι αυτοί που έχουν πανεπιστημιακά πτυχία τείνουν να αποφεύγουν ε, να αναλαμβάνουν εργασίες οι οποίες είναι σε άμεση επαφή με τον ασθενή, δηλαδή με την έννοια ότι του προσφέρουν άμεσες υπηρεσίες με σωματική επαφή μαζί του. Πέστε μας κάντε μια συγκριτική μελέτη, ρωτήστε του ασθενεί στη Γερμανία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία κτλ. που έχουν εξυπηρετηθεί καλύτερα και μετά έλατε να μα πείτε. Η κυρία Ρέιμερς. Εγώ θα μιλήσω για τις γλωσσικές απαιτήσει λόγω και μιας υπόθεσης που εμφανίστηκε στη δική μου εκλογική περιφέρεια. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν γλωσσικές απαιτήσει απέναντι στους νοσηλευτές, αλλά πρέπει να αποφύγουμε και οποιαδήποτε διάκριση από υπερβολές. Πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η δυνατότητα συνεννόησης, αλλά πρέπει να είναι δυνατή και η κινητικότητα μέσα στην Ευρώπη γιατί στη Γερμανία, τουλάχιστον στη δική μου εκλογική περιφέρεια, αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλο έλλειμμα ε, νοσηλευτών και κυρίως ανθρώπων που φροντίζουν ηλικιωμένους. Ενώ στην Ισπανία υπάρχουν, για παράδειγμα, πάρα πολλοί άνθρωποι με ειδικέ γνώσεις και θα μπορούσαν να εργαστούν σε εμά. Έχουμε βάλει λοιπόν ε, Ισπανούς νοσηλευτές οι οποίοι έγιναν πολύ καλά δεκτοί, οι ε, ηλικιωμένοι ήταν πολύ ικανοποιημένοι οι οικογένειε ήταν ικανοποιημένε, ακόμα και οι ίδιοι οι συνάδελφοί του είπαν Μα αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν πολύ καλά. Και τώρα ξαφνικά ερχόμαστε και επιβάλλουμε γλωσσικέ απαιτήσει που θα οδηγήσουν σε απαγόρευση άσκηση του επαγγελματό του. Αυτό είναι στην πραγματικότητα απολύτω αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Που αυτό που θέλουμε είναι κινητικότητα των επαγγελματιών, Θέλουμε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους εκεί ε, που, που βρίσκονται σε χώρες που έχουν υψηλή ανεργία να μπορέσουν να μετακινηθούν σε άλλες χώρες μέλη για να βρουν δουλειά. Εάν τώρα επιβάλλουμε πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια, στενέψουμε δηλαδή τα περάσματα, τις διόδους, τότε πετυχαίνουμε ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή ότι οι άνθρωποι αποστρέφουν πια απογοητευμένοι το πρόσωπό τους από την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ε, εξαντλήσαμε και τον κατάλογο των εγγεγραμμένων. Θα λάβετε αμέσω το λόγο, κυρία μου. Ακούγοντα ωστόσο τις παρεμβάσεις, είδα ότι η γενική σχολική εκπαίδευση έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αν εξετάσουμε τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεργία των νέων μέχρι 50% σε ορισμένες χώρες και σε χώρες μέλη όπου η γενική σχολική εκπαίδευση για να μπορέσει μετά να προχωρήσει σε επαγγελματική εκπαίδευση, η ανεργία είναι στο 8%. Λοιπόν, έχει καλή πρόθεση η πρόταση. Είναι καλών προθέσεων. Για να διαμορφωθούν οι σπουδέ έτσι ώστε να έχουν τη βέλτιστη δυνατή απόδοση. Αν όμω δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το, την τεράστια απίση κόστου, θα Έχουμε ως αποτέλεσμα, φοβούμε, ότι θα έχουμε, αν δηλαδή ισχύσει η εκπαίδευση αυτή, θα έχουμε πάρα πολύ καλά εκπαιδευμένους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες και μετά θα χρειαστεί να φτιάξουμε ειδικά προγράμματα για να εξασφαλιστεί μια νέα κατηγορία η οποία βεβαίως θα αμείβεται λιγότερο καλά και αυτή είναι η πραγματικότητα που σημειώνεται στα περιφερειακά νοσοκομεία. Αυτό το ενδεχόμενο δεν έχει ληφθεί με κανένα τρόπο υπόψη στην πρόταση της Κομισιόν. Και γι' αυτό νομίζω ότι όλοι έχουμε ιδιαίτερο συμφέρον να εξετάσουμε προσεκτικά και να συζητήσουμε με τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Ενίας Αγοράς το κείμενο της κυρίας Βάις Κέρμπερ. Δεν έχω λάβει ποτέ Τόσε πολλές επιστολές, τηλεφωνήματα κλπ. όσο για το σχέδιο αυτό από δημάρχους, από ε, οργανώσεις, από ενδιαφερομένους οι οποίοι ανησυχούν πάρα πολύ. Γι' αυτό έχουμε κάθε ενδιαφέρον και συμφέρον να φροντίσουμε ώστε να μην έχουμε μεν καλές προθέσεις αλλά να βγάλουμε εκτός παιχνιδιού ειδικευμένους νοσηλευτές και νοσηλεύτριες οι οποίοι διαθέτουν την απαραίτητη πείρα αλλά δεν ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις, αυτές τις προϋποθέσεις που πάτε να επιβάλλετε. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα συζητήσουμε ξανά με τους συναδέλφους της ΙΜΚΟ. Προθέσεις καλές αλλά μέχρι τώρα έχω πάρα πολύ μεγάλες επιφυλάξεις ό,τι αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Κομισιόν και μάλιστα εσείς κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας, την εισηγήτρια και όλους τους ευρωβουλευτές που πήραν το λόγο. Τα σχόλια είναι πολύ χρήσιμα. Όπως γνωρίζετε, συζητούμε με τα κράτη-μέλη επί του παρόντος την πρόταση αυτή και με εσάς βέβαια. Και όλες οι προτάσεις και τα σχόλιά σας είναι πάρα πολύ χρήσιμα προκειμένου να καταλήξουμε στο κείμενο το οποίο τελικά θα υιοθετηθεί, ελπίζουμε, την επόμενη χρονιά. Εννοείται, στο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου δεν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας. Έχω όμως σημειώσει μερικές και θα προσπαθήσω να αντιδράσω στα όσα ακούσαμε για να σας βοηθήσω στις δικές σας συζητήσεις προκειμένου να καταλήξετε στη δικιά σας γνωμοδότηση. Πρώτα απ' όλα, για τα επαγγελματικά προσόντα. Το πρώτο που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι Θέλουμε να βρούμε έναν τρόπο που να αποδεικνύει τα επαγγελματικά προσόντα. Δεν πρόκειται για μια άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αυτό θα είναι ένα επιπλέον βήμα. Πρόκειται απλώ για την αναγνώριση. Ό,τι και να κάνουμε, είτε την άρρητη άδεια δώσουμε, αυτό είναι αναγνώριση προσόντων, επαγγελματικών προσόντων και όχι άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Δεύτερον, πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Αυτό το επαγγελματικό διαβατήριο θα είναι ένα κλειστό σύστημα. Οι καθυστερήσεις υπάρχουν γιατί ζητάει η μία αρχή περισσότερες λεπτομέρειες από την άλλη αρχή μέχρι τώρα. Ενώ με την κάρτα αυτή που λέμε εμείς θα είναι γνωστές οι καταστάσεις μεταξύ όλων και το IMI θα βοηθάει η χώρα μέλος από όπου προέρχεται ο ενδιαφερόμενος θα δίνει μια πιστοποίηση για το ότι τα έγγραφα, τα διπλώματα κτλ. είναι αυθεντικά αγνήσια. Οπότε οι καθυστερήσεις που υπάρχουν σήμερα δεν θα υπάρχουν πια ακριβώς εξαιτίας αυτού του νέου συστήματος που προτείνουμε. Και γι' αυτό ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μικρότερες προθεσμίες, ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που μετά από ένα χρόνο δεν έχει απαντήσει μια αρχή. Δηλαδή υποβάλλει κάποιος επαγγελματίας ε, αίτηση και δεν υπάρχει καμία αντίθεση για χρόνια από τι αρχέ κάποιου άλλου κράτου μέλους. Λοιπόν, λαμβάνοντα υπόψη ότι το σύστημα θα είναι κλειστό και ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μα όχι μόνο τι αρχέ που εκδίδουν τα επαγγέλματα αλλά και τι επαγγελματικέ αρχέ, γι' αυτό και προτείνουμε μικρέ προθεσμίε. Αντιλαμβανόμαστε συγχρόνω ότι δεν πρέπει να κολλήσουμε σε αυτό και ότι πρέπει στην πράξη να δούμε ποιες θα πρέπει να είναι οι προθεσμίες. Αυτό συνεπώς είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε. Κοιτάμε δηλαδή μήπως αλλάξουμε κάπως τις προθεσμίες για να δώσουμε περισσότερο χρόνο στις αρμόδιες αρχές για να απαντούν ή μήπως υπάρχει μια ε, περίοδος μετά από την οποία υπάρχει διακοπή αν θέλει επιπλέον πληροφορίες κάποια χώρα από μια άλλη. Δεύτερον, η μερική πρόσβαση. Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα αυτό. Και λαμβάνουμε υπόψη μας βέβαια τα σχόλιά σας και τις ανησυχίες σας. Αλλά πρέπει να έχετε υπόψη σας δύο πράγματα για μας. Το άτομο το οποίο μπορεί να επωφεληθεί από αυτή τη μερική πρόσβαση είναι κάποιος ο οποίος έχει πλήρως τα προσόντα στην χώρα καταγωγής του. Και γι' αυτό για όλα τα επαγγέλματα τα οποία καλύπτονται από την αυτόματη αναγνώριση, δεν πιστεύουμε ότι καλύπτονται από τη μερική πρόσβαση, γιατί τότε είναι αντίφαση. Αν υπάρχει αυτόματη αναγνώριση, δεν τη χρειάζεται κανείς την πρόσβαση, τη μερική. Έχει πλήρη πρόσβαση. Εξορισμού. Αυτό δεν το λέμε στην πρότασή μας, αλλά είναι προφανές για μας τουλάχιστον. Όμως, από την άλλη, Λαμβάνουμε υπόψη μας την πρόταση της εισηγήτριας και πρέπει όντως να το διευκρινίσουμε. Τρίτο, γλωσσικές απαιτήσεις. Αυτό είναι πράγματι πολύ σημαντικό. Και καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τις ανησυχίες σας. Αν κοιτάξετε την οδηγία που ισχύει τώρα, υπάρχει υποχρέωση από τον κλάδο να διαθέτει τα απαραίτητα γλωσσικά προσόντα. Δεν λέει όμως το οποιοδήποτε, προκειμένου να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι για το επάγγελμα αυτό προβλέπεται ήδη η υποχρέωση κατάλληλων γλωσσικών γνώσεων. Εμείς υποθέτουμε στην αρχική πρόταση ότι τα κράτη-μέλη ανάλογα με τις δικές τους πρακτικές πρέπει να αποφασίσουν πώς θα ελέγξουν τις γλωσσικές αυτές γνώσεις. Τα κράτη-μέλη πρέπει να το κάνουν. Αντιληφθήκαμε όμως ότι κάποιες χώρες μέλη πήγαν ακόμα πιο μακριά και δεν ε, επέβαλαν τελικά καθόλου εξετάσεις. Άρα η ιδέα πίσω από τη δικιά μας πρόταση είναι ότι τελικά τα κράτη-μέλη είναι σε θέση και πρέπει να ζητούν κάποια εξέταση, να πετούν κάποιο τεστ. Δεν λέμε ότι πρέπει να παραφορτώσουν τον υποψήφιο με προβλήματα, αλλά να υπάρχει κάποιος τρόπος πιστοποίησης. Τώρα για το γλωσσικό καθεστώς. Αν κάποιος θέλει να δουλέψει στη Φλάνδρα βάσει της οδηγίας πρέπει να διαθέτει τα γλωσσικά προσόντα για να ασκήσει στην ε, περιφέρεια αυτή το επάγγελμά του. Άρα πρέπει να μιλάει Ολλανδικά, Φλαμανδικά τέλος πάντων. Είναι προφανές για μας. Δεν μπορεί να πει, ναι εγώ πρέπει να πάω να δουλέψω στη Φλάνδρα, αλλά μιλάω να, Γαλλικά και Γερμανικά και Γερμανικά θα με εξετάσουν. Ε όχι δεν έχει νόημα αυτό. Συνεπώς για μας είναι προφανές. Από την άλλη, υπάρχει και αναλογικότητα. Αν κάποιος θέλει να δουλέψει στη Φλάνδρα, μπορούμε να πετήσουμε από αυτόν να μιλάει και γαλλικά και γερμανικά, αν δεν θέλει να πάει σε γαλλόφωνη περιοχή, στη Βαλονία ας πούμε. Εδώ πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία. Και ευχαρίστω να συνεργαστούμε με τα μέλη της Επιτροπής σας για να κάνουμε την τελική σωστή πρόταση για τις γλωσσικές απαιτήσει. Για την προειδοποίηση και εδώ υπάρχει για το μηχανισμό προειδοποίησης, υπάρχουν οι σχετικές διατάξεις στην πρότασή μας. Προσπαθώ εδώ να σας πω ότι υπάρχει και στην οδηγία σχετική διάταξη, όχι μόνο ε, στην αρχή στο προημίο. Τώρα για τα επαγγέλματα στα οποία αναφερθήκαμε εδώ, τους γιατρούς γιατί προτείνουμε 5 χρόνια αντί για 6. Αν δείτε την ε, σημερινή οδηγία, λέει 6 χρόνια ή 5.500 ώρες. Τώρα, στις περισσότερες χώρες μέλη ισχύουν και τα δύο. Και τα 6 χρόνια και οι 5.500 ώρες. Αλλά μια-δυο χώρες μέλη το πήραν κατά γράμμα και έχουν 5 χρόνια σπουδές και 5.500 ώρες. Τι θέλουμε λοιπόν εμείς να κάνουμε εδώ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι είναι σαφές πως οι σπουδές αυτές καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας. Όμως, αντιλαμβανόμαστε αυτά που αναφέρατε εσείς εδώ σήμερα και να ξέρετε ότι τα συζητάμε και ευχαρίστως να τα συζητήσουμε παρετέρω και μαζί σας. Έρχομαι τώρα στο τελευταίο θέμα ή νοσοκόμοι. Είναι κάτι που το συζητήσαμε διμερώς με πολλά μέλη της Επιτροπής σας. Τελικά νομίζω ότι διαπιστώνουμε πως μπορεί να υπάρξει ένας συμβιβασμός αποδεκτός από όλους. Αλλά θέλω να σας πω γιατί είναι η πρότασή μας αυτή που είναι. Δεν είναι θέμα κατάρτισης σπουδών, αν προτιμάμε πανεπιστημιακές σπουδές ή όχι. Είναι θέμα οριμότητας. Γι' αυτό και λέμε ότι χρειαζόμαστε άτομα με οριμότητα για να προσφέρουν υπηρεσίες υγείας, μια που υπηρεσίες υγείας γίνονται όλο και πιο περίπλοκες. Μην ξεχνάτε όμως ότι λέμε 12 χρόνια ή αντίστοιχο, ισοδύναμο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το λέτε. Εμείς δεν λέμε 12 χρόνια τελεία και παύλα, λέμε 12 χρόνια ή κάτι που προσφέρει κάτι ισοδύναμο. Μπορεί να είναι δηλαδή 10 χρόνια στο σχολείο συν κάτι ισοδύναμο. Άρα το θέμα δεν είναι κατά πόσο κάνουν καλές ή κακές σπουδές, είναι άλλο το ζήτημα. Και ποτέ δεν υπήρξε η πρόταση του κατά πόσο η επαγγελματική κατάρτιση είναι καλύτερη ή χειρότερη από την ακαδημαϊκή. Αυτό είναι θέμα των χωρών μελών να το αποφασίσουν. Γνωρίζουμε, όπως σας είπα, ποιες είναι οι ανησυχίες σας πάντως. Θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση. Απλώς σας εξηγώ τώρα ποια είναι η προέλευση. Από πού απορρέει η πρότασή μας αυτή. Και μάλιστα μετά από συζητήσεις που είχαμε με τους ενδιαφερόμενους και με τους νοσοκόμους. Να σας ενημερώσω επίσης ότι πρόσφατα ε, κάποιος κλάδος νοσοκόμων ήρθε σε επαφή μαζί μας που μας έδωσε ένα κατάλογο με αρμοδιότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε κάποιο άρθρο. Θα το συζητήσουμε και μαζί σας αυτό πάντως. Εν προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συμβασμό αποδεκτό και από σας και από μας που σημαίνει ότι θέλουμε να συμφωνείτε και σας και να μην το φορέσουμε στενό κορσέ σε κανένα. Και να φροντίσουμε φυσικά να υπάρχει κατάλληλη κατάρτιση για τους νοσοκόμους. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος κ. Γκρότη, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχετε προκαλέσει ορισμένες συναδέλφους να ξαναλάβουν το λόγο. Έχουμε ξεπεράσει κάθε όριο βέβαια του χρονοδιαγράμματός μας. Θα δώσω πάλι το λόγο στην εισηγήτρια και βέβαια θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ λέει κυρία Βάης Κέρμπερ. Ευχαριστώ πρώτα για την συζήτηση που έγινε με τους συναδέλφους μου και ευχαριστώ ιδίως την κυρία Ροτ Μπέρεντ τον κύριο Γκρότε, αλλά και τους άλλους συναδέλφους που έθεσαν το θέμα των ε, νοσηλευτριών. Το κατασκευαστικό σφάλμα, θέλετε, της Κομισιόν είναι ότι επιθυμεί να βελτιώσει την εκπαίδευση των νοσηλευτριών. Δεν ασχολείται όμως με το περιεχόμενο της ειδική εκπαίδευσης των νοσηλευτριών, παρά μόνο με το επίπεδο της σχολικής εκπαίδευσης που χαίρουν σε κάθε χώρα μέλος όπου για παράδειγμα στη Μεγάλη Βρετανία έγινε πανεπιστημιακές, έγιναν πανεπιστημιακές οι ε, σπουδές αυτές, εν τέλει όμως είναι λιγότερο καλά τα προσόντα που διαθέτουν οι νοσηλεύτριες. Πρέπει λοιπόν να εξεταστούν οι περιπτώσεις των χωρών εκείνες, εκείνων οι οποίες έχουν αυτή την διπλή ε, εκπαίδευση και που έχουν εξασφαλίσει πολύ υψηλό επίπεδο προσφερωμένων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί η αντιστοιχία, αντιστοιχία με τα 12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης που εξασφαλίζεται από το περιεχόμενο των σπουδών και την υψηλή ποιότητα των σπουδών των νοσηλευτριών. Γι' αυτό θα ε, με ικανοποιήσει ιδιαίτερα αν δεχτείτε την πρόταση που κάνω εγώ. Έχω και μια παράκληση, γιατί η κυρία Ροτ Μπέρεν σωστά είπε ότι πρέπει να μιλήσουμε με την ΙΜΚΟ, την κυρία Βερνιού και άλλους συναδέλφους και θα ήταν πολύ καλά να έχουμε μια ξεκάθαρη θέση δική μας για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε συνολικά την πρόταση της Κομισιόν. Τώρα, πολύ σύντομα για τα γλωσσικά, για τις γλωσσικές απαιτήσει. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει η κυρία Μπρέπολς. Από την άλλη, ακούω και την κυρία Γιανακουδάκη που λέει ότι δεν πρέπει να ξεφύγουμε από την αναλογικότητα. Ίσως το σωστό είναι να ακολουθήσουμε την μέση οδό, να πούμε δηλαδή ότι σε περιπτώσεις χωρών με πολλές γλώσσες, όπως για παράδειγμα η Φλάνδρα, στο Βέλγιο πρέπει να μπορεί ο εργαζόμενος ή αυτό που επιθυμεί να εργαστεί να μιλάει την γλώσσα που κυρίω μιλείται εκεί. Τώρα για το επαγγελματικό διαβατήριο και η Κομισιόν λέει οικειοθελώ. Εγώ ε, υποστηρίζω βέβαια αυτό, είμαι γενικά υπέρ του εθελοντικού χαρακτήρα, αλλά είμαι ανοιχτή στη συζήτηση. Πρόσβαση στον ασθενή. Κυρίω εκεί πρέπει να παίξει ρόλο το κριτήριο τη ασφάλεια του ασθενού και βέβαια πρέπει να είναι υψηλέ οι απαιτήσει. Βέβαια και εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για την κατάσταση των Πολωνών. Είμαι ανοιχτή κυρία Χίπνερ γιατί γνωρίζω ότι στην Πολωνία πράγματι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά τα τελευταία χρόνια. Εκπληρούνται οι προϋποθέσεις. Για τον κύριο Πυρίλο για την ε, κατεξουσιοδότηση πράξη ας μην ότι η Κομισιόν με τις κατεξουσιοδότηση πράξης έχει αυξήσει τις δυνατότητές της να τροποποιεί τις οδηγίες. Και εφόσον εμείς συμμετέχουμε ως Κοινοβούλιο, γνωρίζετε άλλωστε πόσο γρήγορα επεξεργάζονται τις ε, ε πράξη, πόσο γρήγορα προχωρούν δηλαδή, είναι σημαντικό καμιά φορά να συμμετέχουν, δηλαδή να συμφωνεί κανείς και με τις χώρες μέλη. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα πράγματα λίγο πιο διαφοροποιημένα και για τις προθεσμίες εν τέλει και εγώ τάσομαι υπέρ των συντομότερων προθεσμιών απέναντι στο status αλλά θεωρώ ότι οι προθεσμίε που προτείνει η Κομισιόν είναι πάρα πολύ περιορισμένε, πολύ σύντομε. Τώρα, για τι γλώσσε, επανέρχομαι. Δέχομαι και το επιχείρημα της Γερμανίδας συναδέλφου της FDP, της φιλελεύθερης δηλαδή, που λέει ότι δεν πρέπει να περιορίσουμε την ε, κινητικότητα με κανέναν τρόπο. Αλλά βέβαια Γλώσσες είναι γλώσσες. Ε, νομίζω ότι μπόρεσα να απαντήσω σε λίγο πολύ όλα τα ερωτήματα. Ευχαριστώ κύριε Βαϊσκέρβερ και προθεσμία κατάθεση τροπολογιών είναι 8 Δεκάτου. 6 Νοεμβρίου ψηφοφορία, εδώ δηλαδή, και στην ΙΜΚΟ γίνεται η ψηφοφορία στις 28 Νοεμβρίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Θα δούμε τώρα πώς θα προχωρήσουμε. Κατά τα άλλα το επόμενο θέμα είναι η έκθεση Αρσένη, το υπαριθμό 19. Το λόγο έχει αμέσως ο εισηγητής. Thank you, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, μια που 326 τροπολογίες είχαμε συνολικά. Η έκθεση αυτή είναι τεχνικού χαρακτήρα, οπότε πραγματικά έχουν κάνει εκπληκτική δουλειά για να έχουν καταθέσει τόσες τροπολογίες. Βέβαια, πολλοί προσπάθησαν ε, να καταλάβουν ε, τις τεχνικές πτυχές, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές. Πάντως να έχετε υπόψη σας ότι όσο μπορούν να σας βοηθήσουν οι υπηρεσίες μου στο τεχνικό σκέλος, ευχαρίστως να το κάνουμε. Ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να τις υποβάλλετε. Όντω λοιπόν είναι πολύ τεχνική αυτή η έκθεση. Συγχρόνω όμως, από πίσω υπάρχει και ένα τεράστιο πολιτικό ζήτημα. Στον Ντέρβαν αποφασίσαμε για το LULUCF, για την χρήση γης, αλλαγές χρήσης γης και δοσοκομεία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να μεταφέρει τη συμφωνία αυτή, την απόφαση αυτή, να την κάνει κοινοτικό και εκτιμένο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα πολύ καλό μήνυμα, ότι δηλαδή τιμούμε την υπογραφή μας στις διαπραγματεύσεις και όντως έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προχωρήσουμε με την εφαρμογή της απόφασης αυτής. Και υπάρχει συνένεση για το ότι ό,τι συμφωνήθηκε μέχρι τώρα στο Τέρμαν μπορεί εύκολα να γίνει κοινοτικό και εκτιμένο. Αυτό το αποφασίσαμε μετά από διαβούλευση με τις χώρες μέλη. Αυτό όμως που αντιμετωπίζουμε σήμερα πάει ακόμα πιο πέρα. Το θέμα που μας απασχολεί όμως είναι ένας άλλος στόχος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, δεν το καθένα, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, μπορεί να εξοικονομήσει πάρα πολλά από την ε, μείωση των ε, εκπομπών από τη χρήση γης, τις αλλαγές χρήσης γης, τη δασοκομεία, από τους υγρότοπους κλπ. Είναι οι οικονομίες που δεν ε, γίνονται αισθητέ από τους πολίτες μας στις χώρες μας, δεν τις αντιλαμβάνονται έτσι από πρώτο χέρι. Και γι' αυτό λοιπόν με την πρόταση αυτή υπάρχουν τρία πράγματα που έχουμε συμπεριλάβει. Το ένα είναι η λογιστική καταχώρηση από τις αγροτικές δραστηριότητες και ξέρετε ότι εδώ πέρα βάζουμε και την αποστράγγιση και την επανήγρανση των ε, υγροτόπων. Θέλουμε τη συνοχή και θέλουμε επίσης και τη δυνατότητα αναγνώρισης ώστε να μπορούν να γίνονται τεχνικές ε, προσαρμογές στα σημεία αναφοράς. Αυτά τα τρία λοιπόν νέα ζητήματα που έχουν να κάνουν την απόφαση του Ντέρμπαν, δεν συζητάμε εδώ βέβαια ακριβώ για τη χρήση γης αλλαγή, χρήση και δασοκομεία, αποτελεί και την προετοιμασία που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να περάσει σε ένα δεύτερο στάδιο όπου γίνεται και η λογιστική καταχώρηση των Λούλουσεφ και άρα οι οικονομίες που κάνουμε από την μείωση προσπάθειας που γίνεται για την μείωση των βιομηχανικών ε, εκπομπών. Προσθέτουμε σε αυτές δηλαδή και τις γεωργικές, καταλογίζοντας τις κανονικά. Και το κάνουμε και πιο σωστά, γιατί λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις εκπομπές. Και άρα λαμβάνουμε υπόψη μας και τις κρυφές οικονομίες που κάνουμε, οι οποίες μέχρι τώρα δεν καταλογιζόντουσαν. Προκειμένου λοιπόν να φτάσουμε σε ένα επίπεδο όπου να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την οικονομία μειώνοντας τις βιομηχανικές μας εκπομπές, πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο συνοχής, όπως ακριβώς έχουμε με τις βιομηχανικές εκπομπές και να το κάνουμε αυτό και εδώ και σε αυτό το τομέα. Αν λοιπόν θέλουμε τώρα να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο και να μειώσουμε τις εκπομπές μας ε, από τη χρήση γης κλπ, τι πρέπει να κάνουμε. Η Δανία, η Ισπανία και η Πορτογαλία υπολογίζουν ε, τις οικονομίες εκπομπών από τις αγροτικές εκπομπές, ενώ άλλες χώρες δεν μετράνε τις οικονομίες που κάνουν εκείνοι στον αντίστοιχο τομέα. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι εδώ, σε αυτή την αίθουσα, θα τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Γιατί? Γιατί δεν ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Γιατί άλλοι κάνουν περισσότερες προσπάθειες από άλλους και άλλοι τις υπολογίζουν αυτές τις προσπάθειες που κάνουν, ενώ άλλοι που τις κάνουν δεν μπορούν να τις υπολογίσουν. Άρα τίθεται θέμα ανταγωνισμού τελικά. του ανταγωνισμού μεταξύ των 27 μας χωρών. Γι' αυτό, λοιπόν, αν θέλουμε να περάσουμε στο δεύτερο στάδιο, δηλαδή να υπολογίζουμε και τις οικονομίες αυτές που γίνονται στις εκπομπές από την χρήση γης, αλλαγές χρήση και δοσοκομείας, τότε πρέπει σε αυτή την νομοθεσία που αποφασίζουμε τώρα να συμπεριλάβουμε τις τρεις αρχές. Και αυτό θα υποστηρίξω, ότι δηλαδή όλοι υπολογίζουμε τα ίδια πράγματα με τον ίδιο τρόπο και ότι έχουμε και τρόπο μεταξύ μας να ενημερώνουμε ένα τον άλλον για το τι κάνουμε και έτσι να διδαχτούμε και από τις βέλτιστες πρακτικές. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δηλαδή δεν υπολογίζουμε τέτοια πράγματα με τον ίδιο τρόπο και δεν ενημερώνουμε ένα τον άλλον για το τι κάνουμε, ας ξεχάσουμε το δεύτερο στάδιο. Ας αποφασίσουμε ότι δεν θα περάσουμε στο στάδιο συμπερίληψης και των LULUCF. E Είχαμε μία ακρόαση πριν από λίγες μέρες για αυτό το θέμα και ευχαριστώ και τους συναδέλφους που παρευρέθηκαν εκεί. Εκεί λοιπόν καταφέραμε δύο μύθους του Ντέρμαν να τους καταρρύψουμε. Ο πρώτος μύθος και μάλιστα ήταν ο πρόεδρος του Πεκαγέγα από την Ένωση των Γεωργών που μας βοήθησε σε αυτό. Είναι ότι υπάρχει γραφειοκρατία μεγάλη για τους ε, Γιώργους. Οι ίδιοι δηλαδή, οι επικεφαλής των λόμπι που εκφράζουν τα συμφέροντα του γεωργικού κόσμου δηλαδή μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πρόεδρος είπε ότι σε αυτή την νομοθεσία εδώ που συζητάμε τώρα δεν υπάρχει γραφειοκρατία και βάρος για τους γεωργούς. Ο ίδιο το είπε. Και ο πρόσωπος του GRC επίσης είπε ότι εδώ μιλάμε για μια άσκηση που θα γίνει σε μακροστατιστικό επίπεδο. Δεν θα γίνει ατομικά με εγκαταστάσεις ανά γεωργική εκμετάλλευση. Θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία τα οποία ήδη δίνουν τα κράτη-μέλη, UNFT των ΗΕ, δηλαδή την υπηρεσία, και στη Κυβερνητική Επιτροπή δηλαδή για την αλλαγή του κλίματος. Θα παίρνουμε στοιχεία λοιπόν και από εκεί. Ο δεύτερος μύθος που καταλήφθηκε είναι ότι αυτή η νομοθετική πρόταση ε, πλήττει τα κυρίαρχα δικαιώματα των χωρών. Και αυτό είναι μύθος. Δεν ισχύει. Έχω διαβάσει λεπτομερώς και έχω κατανοήσει το έγγραφο. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν ότι από τη δικιά μου την πλευρά θα λέγεται σαφώς ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο με αυτή την νομοθετική πρόταση. Έχουμε λοιπόν τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Σας διαβεβαιώνω λοιπόν δεν υπάρχει ούτε γραφειοκρατία ούτε θέμα εθνικής κυριαρχίας με την νομοθετική αυτή πρόταση. Θα μείνω λοιπόν στις αρχές αυτές και θέλω να ακούσω και τις δικές σας σκέψεις και προτάσεις. Και επαναλαμβάνω ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου είμαστε στην διάθεσή σας. Ό,τι τεχνικές επεξηγήσεις θέλετε, ό,τι πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Μη διστάσετε. Θέλω, ακόμα και αν δεν περάσει με πλειοψηφία αυτή η πρόταση, τουλάχιστον να περάσει συναντικά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τους κοιόδης συζητητές, ο κύριος Ζίμπερ. Ε, ε, Ο Ζέμπερ, ε, ευχαριστώ. Η συνάδελφό μας που είναι σκιώδη ε, δεν ε, σήμερα, δεν μπορεί να είναι παρούσα και γι' αυτό με παρακάλεσε να τα πω εγώ. Ευχαριστούμε τον Κρήτονα για την εργασία του και έχουμε πλήρη κατανόηση για την επιθυμία της Κομισιόν που θέλει να φτιάξει μια καλύτερη βάση για την κλιματολογική μας πολιτική. Βέβαια, ο τομέας αυτός παράγει, προκειμένου δηλαδή, 9% των αερίων θερμοκηπίου. Βέβαια, δεν είναι τέλειοι οι κανόνες, ούτε τέλεια η τράπεζα δεδομένων, η βάση δεδομένων, αν και σε άλλους τομείς υπάρχουν ακόμα λιγότερα δεδομένα. Η δική μας βασική ανησυχία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και οι διάφορες παρεμβάσεις του κ. Μέτσκερ, Διευθυντού της Κομισιόν, δεν μας επέτρεψαν να ξεπεράσουμε, ας πούμε, τις ε, ανησυχίες μας αυτές. Οι ανησυχίες μας είναι ότι και χώρες μέλη από τη μια μεριά, αλλά και ολόκληρο ο γεωργικός τομέας από την άλλη μεριά, θα δουν να τους επιβάλλονται κάποιες επιβαρύνσεις, δηλαδή συλλογή δεδομένων, υποβολή ε, εκθέσεων ή αναφορών κλπ. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να τηρήσουμε τα διεθνώς συμφωνημένα, δηλαδή στα πλαίσια της ε, διάσκεψης του κλίματος των Ηνωμένων Εθνών και του πρωτοκόλου του Κιώτο και να προσπαθήσουμε, ίσως και με την υποστήριξη της Κομισιόν, να φτάσουμε σε μια κοινή μορφή διαβίβασης μεταξύ των χωρών μελών και έτσι να υποστηρίξουμε τις χώρες μέλη διότι εν τέλει η υπόθεση της κοινή αγροτική πολιτικής ίσω υποφέρει και από υπερβολική ρύθμιση. Οποιεδήποτε περαιτέρω υποχρώσεις, έστω και αν στατιστικά έχουν σημασία, κατά τη γνώμη μας δεν είναι σκόπιμε, τουλάχιστον στην παρούσα χρονική περίοδο. Και δεν θα συμφωνήσουμε κιόλα. Οι γεωργοί μα πρέπει να μείνουν γεωργοί, αγρότε. και όχι να αναλάβουν ακόμα παραπάνω καθήκοντα. Έχουμε την παράκληση να εξεταστεί η εφαρμοσιμότητα των προτάσεων αυτών. Μόνο και μόνο με το ότι θα έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα δεδομένα δεν σημαίνει ότι θα προστατεύσουμε καλύτερα το κλίμα. Νομίζω ότι με άλλους τρόπους μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Πρέπει να δούμε αν και πραγματικά όλος αυτός ο όγκος δεδομένων που καταλήγουν εδώ στις Βρυξέλλες όντως συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας καλύτερης πολιτικής. Εξετάζοντας την διεθνή κατάσταση βλέπουμε ότι εξακολουθούμε να είμαστε πρωτοπόροι και καλά κάνουμε. Απλώς ζητώ συγγνώμη αλλά θεωρούμε ότι οι εγγυήσει που δίνονται δεν είναι επαρκείς. Δεν θέλουμε περισσότερες επιβαρύνσεις ούτε για τις χώρες μέλη ούτε για την γεωργία. Τηρούμε τις υποσχέσεις που έχουμε δώσει διεθνώς αλλά νομίζω παραπέρα δεν θα υποστηρίξουμε πολιτικά τίποτα. Ευχαριστώ κύριε Ζέμπερ. η σκιώδης εισηγήτρια των φιλελευθέρων που επίσης εκπροσωπείται σήμερα. Ναι, εκπροσωπώ την κυρία Μάνερς και έχουμε καταθέσει και εμείς τροπολογίες για να επιμείνουμε στην εθελοντική βάση εφόσον υπερβαίνει τα συμφωνημένα στο Τέρμπαν. Υποστηρίζουμε βέβαια το σχέδιο του Ντέρμπαν και θεωρούμε ότι πρέπει προς αυτήν την κατεύθυνση να κινηθούμε και στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά νομίζουμε ότι υπερβαίνουν τα όρια κάποιες υποχρεώσεις που πάνε να επιβληθούν ακόμα στις ε, χώρες μέλη. Διότι αφενός πράγματι η δασοκομική πολιτική εξακολουθεί να ε, υπάγεται στην επικουρικότητα των χωρών μελών και από την άλλη μεριά στην Γεωργία ήδη γίνεται συλλογή τεράστιων όγκων δεδομένων στον γενικό αγροτικό τομέα. Και εγώ προσωπικά έχω να προσθέσω ότι διαπιστώνουμε ότι αυτή η μεγάλη συλλογή ε, των δεδομένων έχει ως συνέπεια μόνο διόγκωση των υπηρεσιών της Κομισιόν και διόγκωση των δαπανών. Το ζήτημα είναι εφόσον συλλέγονται δεδομένα να τα επεξεργάζονται κιόλα κάποιοι και να εξάγουν συμπεράσματα. Εγώ διαπιστώνω από την εμπειρία μου ως αγρότησα ότι κάθε νέο κύμα συλλογής δεδομένων που επιβάλλεται στις χώρες μέλη καταλήγει στο τέλος ε, να φορτώνεται στους ώμους του αγρότη που ο αγρότης στο κάτω της γραφής έχει καθήκον είτε να παράγει ε, τρόφιμα είτε να παράγει εσοδίες οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία καυσίμου κτλ. Αλλά όχι να περνάει όλο τον υπόλοιπο χρόνο του με γραφειοκρατικές υποχρεώσεις. Πρόκειται για υπερβολική επιβάρυνση ενός επαγγελματικού τομέα που οδηγεί και σε μεγάλη απογοήτευση απέναντι στην Ευρώπη. Έχοντας λοιπόν πει αυτά, σημειώνω επίσης ότι αναμένουμε με ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση και σίγουρα πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βρούμε ένα συμβαστικό δρόμο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά του, για τις ενημερώσεις που είχαμε, για την ακρόαση που κάναμε. Με ενδιαφέρον ακούω αυτά που λέω. Ελπίζω να φτάσουμε σε συμβιβασμό, αλλά βλέπω ότι ο καθένα είναι προσκολλημένο μέχρι στιγμή στην άποψή του. Ελπίζω να υπάρξει μια μετακίνηση, γιατί αλλιώ ο συμβιβασμό θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Από τα επιχειρήματα που ακούω, εκπλήσωμαι ακόμα λίγο. Καταρχά, μιλάμε για την λογιστική καταχώρηση για του βοσκότοπου και τη γεωργική γη. Ε, ακούω ε, τους συναδέλφους που λένε δύσκολο να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Διαβάστε την έκθεση IPCC. Υπάρχουν ούτως ή άλλως πάρα πολλά από αυτά τα δεδομένα για κάθε κρατός μέλος. Υπάρχουν τα δεδομένα. Υπάρχουν πολλές δορυφορικές πληροφορίες. Όλες αυτές οι πληροφορίες ε, για τις εκπομπές υπάρχουν ε, για τις εκπομπές. Υπάρχουν ε, δεδομένα Τώρα, για το αν θα βαρύνει πολύ αυτό το μεμονωμένο γεωργό, αυτό το επιχείρημα δεν με πείθει, αφού υπάρχουν αυτά τα δεδομένα. Πάμε στον Ντέρμπαν και στη συμφωνία Ντέρμπαν. Στον Ντέρμπαν δεν συμφωνήσαμε ότι είναι υποχρεωτική αυτή η λογιστική καταχώρηση. Παρ' όλα αυτά, ζητάμε από τις αναπτυσσόμενες χώρες όταν συμμετέχουν να καταχωρίζουν όλοι, όλες τις εκπομπές από την χρήση γης και αλλαγή χρήση γης. Μετά από το 2020, ούτως ή άλλως το 2015 θέλουμε να έχουμε μια κλιματική συμφωνία και η Ευρώπη διεθνώς θα υποχρεωμένη να δίνει στοιχεία. Γιατί τα ζητάμε ήδη από τις ανεπτυγμένες χώρες τώρα και οι ανεπτυγμένες χώρες είναι σίγουρο ότι θα ζητήσουν την ίδια προσπάθεια και από τις ανεπτυγμένες χώρες δεν πρέπει να περιμένουμε, ή μάλλον μπορούμε να περιμένουμε, αν θέλετε, μέχρι το 2020, μέχρι να μας υποχρεώσουν το κάνουμε, ή να είμαστε συντονισμένοι εκ των προτέρων. Αλλά προ αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε. Υπάρχουν τα δεδομένα διεθνώς, τα ζητάμε από τις αντισώμενες χώρες, αν, ε, συμμετάσχουν στο, συμμετέχουν ήδη στο Red Plus, και θα χρειαστεί να το κάνουμε και οι ίδιοι. Τώρα, για το σχέδιο δράση που είναι τμήμα τη πρόταση. Και εδώ συνειδητοποιούμε ότι το λουλουσιέφ συνολικά είναι υπεύθυνο για το 17% των ε, εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Με βάση τους μακροπρόθεσμους στόχους μας ξέρουμε ότι και ο τομέας LULUCF θα πρέπει να βοηθήσει στη μείωση. Ε, ξεκινάμε τώρα με σχέδια δράσης όπου τα κράτη-μέλη, του ζητάμε ευγενικά, τουλάχιστον να μας δώσουν κάποιες προφορίες για το προς τα που κατευθύνονται δεν είναι και τόσο φιλόδοξη δά η πρόταση τη Κομισιόν, τόσο υπερβολική. Και εγώ μάλιστα προτείνω και τροπολογίε ούτω ώστε να γίνει πιο φιλόδοξη. Δηλαδή ε, να έχουμε και στόχου στο Λουσιεφ, γιατί αλλιώ ποτέ θα πετύχουμε τη μείωση που θέλουμε. Δύο μικρά ε, θέματα τα οποία δεν έχουν αναφερθεί, γιατί συζητάμε συνέχεια το σχέδιο δράση τη Λουλουσιεφ και τα ε, υποχρεωτικά στοιχεία για του τους και τις, ε, την καλλιεργήσιμη γη. Ε, αυτή είναι μια πολιτική συζήτηση. Ελπίζω λοιπόν να, να γίνει η πρόοδος, θα είναι δύσκολο να αποφύγουμε την διπλωμε... καταχώρηση για τη βιομάζα. Θα πρέπει στη λογιστική καταχώρηση οι εκπομπές της βιομάζας, γιατί αν κόψεις ένα δάσος θα υπάρξουν εκπομπές, να πρέπει να καταχωρούνται στο LULUCF. Για τους υγρότοπους τώρα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα σημαντικό τομέα. Ε, προκαλούνται πολλέ εκπομπέ, κυρίω μεθανίου εδώ. Μπορείτε να πείτε ότι η δεύτερη, ο δεύτερος μεγαλύτερο εκπομπός τέτοιων αερίων είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως θα πρέπει να λογαριάζουμε και τις εκπομπές των υγροτόπων. Δεν έχουμε υποχρεωτικά, υποχρεω διεθνή δέσμευση τώρα, διεθνή υποχρέωση, αλλά ας αρχίσουμε από τώρα, ούτω ώστε τα δεδομένα που θα δίνουμε στη γραμματεία του UNFCCC να είναι σωστά, λογικά, αξιόπιστα. Αυτό προσπαθεί να πετύχει αυτή η πρόταση. Σας παρακαλώ, τέτοια επιχείρηματα θέλω να ακούσω, παρά να λέμε «Α, δεν μπορώ, τέλο πάντων, τη γραφειοκρατία» κτλ. Ε, αυτά δεν, δεν στέκουν, αυτά τα επιχείρηματα περί υπερβολικής γραφειοκρατίας. Η äh, κυρία Ρόσπαχ, που εκπροσωπεί την της Ιούδια. Ευχαριστώ. Αντικαθιστώ την Τζούλη Γκέρλι. Θα προσπαθήσω να σας πω εγώ τι ήθελε να σας πει. Να κάνω και μία μικρή μετά προσωπική παρατήρηση. Ξέρετε ότι εδώ στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συχνά δημιουργούμε ουτοπιστικούς κανόνες, ε, φιλόδοξους στόχους, υπερβολικούς για τους γεωργούς. Σας παραπέμπω σε αυτά που είπαν συνάδελφοι Γερμανοί πριν από λίγο. Αυτή η υποχρέωση κοινοποίηση για την λογιστική καταχώρηση, για την καλλιεργήσιμη γη και τους βοσκότοπους είναι κανόνες ανέφικτοι, ουτοπιστικοί. Τι να πω, πρέπει να το επαναλάβω κι εγώ, συμφωνώ απόλυτα. Τώρα, για αυτά που θέλει να πει η Τζούλι Καταρχάς, να ευχαριστήσουμε την Κομισιόν και κυρίω τον Κρήτονα Αρσένη για την έκθεσή του. Φυσικά ένα σημαντικό θέμα που μας ξαναφέρνει μπροστά στις ευθύνες μας σε ό,τι αφορά τη γεωργική πολιτική. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες για την έκθεση, γιατί θεωρούμε ότι η αρχική πρόταση της Κομισιόν και το κείμενο που μας προτείνει ο Κρήτονας πάνε πιο πέρα από τον Τέρμπαν. Νομίζουμε ότι το κείμενο αυτό είναι ουτοπιστικό και υπερβολικά φιλόδοξο και, εν πάση περιπτώσει, μα καταλαμβάνει εξαπίνη. Πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Μα επιβάλλεται πράγματα πολύ γρήγορα. Η χρήση αυτή τη γη θα πρέπει να είναι ένα τμήμα ενός πακέτου διεθνούς. Γιατί αν εμεί τα δεχτούμε όλα αυτά, θα έχουμε ένα άχθος εργασία πολύ μεγαλύτερο από άλλα κράτη που δεν έχουν τι ίδιε υποχρεώσει. Μα αρκεί το άρθρο 10 με τα εθνικά σχέδια. Η Κομισιόν προσπαθεί να μας πείσει για το αντίθετο. Εμεί πιστεύουμε ότι με αυτά που λέτε θα υπάρξει ένα επιπλέον άχθος, το οποίο θα είναι απίστευτα επαχθε. και για τα κράτη-μέλη και για του γεωργού. Θα υπάρξει λοιπόν μια διπλή νομοθεσία. Θα έχει μια λογιστική καταχώρηση του δεύτερου πυλώνα και παράλληλα μια λογιστική καταχώρηση για οικολογικούς σκοπούς, ας πούμε, για το περιβάλλον. Δεν νομίζω ότι τα εθνικά σχέδια θα πρέπει να τροποποιηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Γι' αυτό η σκιώδης συγγήτρια θα κάνει προτάσεις, ούτως ώστε να συμβάλλουμε προς την επίτευξη συμβασμού. Οι τροπολογίες της έχουν σαν στόχο να μειώσουν το βάρος που θα πέσει στα διαφορα ούτω ώστε τα σχέδια δράσης να είναι πιο ευέλικτα και να μειώνεται η παρέμβαση της ε, Κομισιόν. Όταν μιλήσαμε τον Ιούλιο για την ε, πρόταση της Κομισιόν, είχε πει ότι η Κομισιόν πάει υπερβολικά μακριά και για τις κατεξουσιοδότησει πράξεις. Μιλάμε εδώ για πράγματα τα οποία θα πρέπει να ρυθμίζονται με την τακτική νομοθετική διαδικασία και όχι μέσω της επιτροπολογίας. Ευχαριστώ την κυρία Ρόσμπαχ. Ακούσαμε όλους τους κοιόδης συγητές ή τους εκπροσώπους τους. Θα διαβάσω τα ονόματα των υπολείπων που έχουν εγγραφεί. Jolanta Χίπνα, dann die Kollegin Kukovic, dann äh, der Kollege Sadurikakis, Sadurskis, dann der Kollege Prodi, Kollege Μήπως ξέχασα κάποιο όνομα? Όχι. Καλά λοιπόν. Άρα μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στον κατάλογο των εγγεγραμμένων, αλλά για δύο λεπτά ο κάθε ένας ή η κάθε μία. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με τον χρόνο. Και έχουμε μια έκθεση ακόμα για, την, τον θόρυβο των αεροπλάνων. Η κυρία Κλάς, ευχαριστώ. Πράγματι μπορεί κανείς να συζητήσει για ώρες, αλλά πολλά λέχθηκαν ήδη. Και επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο Ρίχαρτ Ζέμπερ και η Άννα Ρόσπαχ. Η διάσκεψη κλίματος στο Ντέρμπαν συμφώνησε ότι θα περιλάβουμε υποχρεωτικά την δασοκομεία από το 2013. Έρχεται τώρα η Κομισιόν και περιλαμβάνει με την πρότασή τη ήδη την δασοκομεία. Άρα πρόκειται για ας πούμε ένα είδος υπερβάλλοντος ζήλου που θα οδηγήσει σε γραφειοκρατία, θα οδηγήσει και σε στρέβλωση του ανταγωνισμού, διότι υπενθυμίζω ότι κάθε δεδομένο που συλλέγεται πρέπει και να γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας. Άρα πράγματι θα υπάρξει μεγαλύτερη γραφειοκρατία. Είναι λάθο να το αμφισβητούμε αυτό. Εξάλλου, το να βάλουμε μέσα και την αγροτική πολιτική και τα εθνικά σχέδια για την διατήρηση των ε, βοσκοτόπων, πάλι αυτά θεωρώ ότι δεν είναι σωστά. Βρισκόμαστε μέσα στα πλαίσια τώρα της μεταρρύθμισης της αγροτικής πολιτικής και αγωνιζόμαστε να πετύχουμε ρεαλιστικούς στόχους. Ας μην αντιβαίνουμε σε αυτούς. Με αυτό το νόημα πρέπει να εξεταστεί και αυτό το screening. Τώρα, για την δασοκομεία. Σωστό είναι που το πρωτόκολλο του κλίματος επεκτείνεται και σε αυτό και στην δασοκομεία. Αφενός, αφενός αυτό αφέτερο, όμως το δάσος πρέπει να εξεταστεί και με την έννοια ότι η βιώσιμη ε, δασοκομεία είναι σημαντικός στόχος και από μόνος του, διότι το δάσος απορροφά διοξίδιο του άνθρακα. Επομένως, μπορεί αυτή η συμβολή του δάσους να εμφανιστεί καλύτερα. Και γνωρίζουμε ότι εάν το δάσος δεν καλλιεργείται, δηλαδή δεν το φροντίζουν, ε, θα αγριέψει και τελικά τα δέντρα κινδυνεύουν να ε, καταστραφούν, να ξεραθούν δηλαδή και ούτω καθεξής. Άρα αυτό είναι σημαντικό. Επίσης ε, εκμετάλλευση του δάσου ό,τι αφορά τη συλλογή τη ξυλία. Και αυτή είναι σημαντική, διότι η ξυλία αυτή χρησιμοποιείται και για καύσιμο. Άρα, εδώ υποστηρίζω εγώ την βιώσιμη εκμετάλλευση του δάσου. Ευχαριστώ, κύριε Χίπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς καμιά αμφιβολία, η χρήση γης και οι αλλαγές στη χρήση γης είναι κάτι πολύ σημαντικό για να υπολογίσουμε τις εκπομπές. Όμως θα μπορούσε κάποιος να κάνει κάπως πιο ήπια την πρόταση αυτή, εφόσον αποφάσιζε να μην γίνονται όλα αυτά σε υποχρεωτική βάση, αλλά σε θελοντική βάση. Όπως είπαν κάποιοι συνάδελφοι στο Ντέρμπαν, δεν υπήρξε υποχρέωση. Είπαμε ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να εισαχθούν και ότι οι χώρες από μόνες τους θα αποφάσιζαν πόσο μακριά θα ήθελαν να πάνε. Η έκθεση του κύριου Αρσένη είναι ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας. Όμως, θέλω να τονίσω κάποιες διατυπώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες είναι προβληματικές για μας. Για παράδειγμα, τα κράτη-μέλη πρέπει να ετοιμάσουν προγράμματα δράσης ε, για τη μείωση των εκπομπών από την αλλαγή χρήση γης. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως πρέπει μετά να τα αλλάξει, να τα τροποποιήσει. Αυτό πρέπει να γίνεται σε θελοντική βάση από τις χώρες-μέλη. Και οι χώρες από μόνες τους θα θέλουν τότε να δείξουν ότι κάνουν πολλά για να μειώσουν τις εκπομπές. Γιατί αν η βιομηχανία ε, προκαλεί εκπομπές ε, και η γεωργία επίσης. Έπειτα, προτείνει κατά εξουδότηση πράξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι σωστό γιατί επηρεάζει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Κάτι άλλο που με απασχολεί είναι οι εκπομπές που έρχονται από τους υγρότοπους ε, και βοσκοτόπους. Και αυτό θα πρέπει να είναι σε θελοντική βάση. Όλοι έχουμε υπογράψει το Κιώτο και ξέρουμε τι είναι η δεσοκομεία. Αν αλλάξουν οι ορισμοί τώρα και αλλάξουν όλα αυτά, αυτό δεν θα ήταν καλό. Ιδιαίτερα όταν σε άλλες μικρές χώρες τα δάση αποτελεί πλούτο της χώρας, όπως στη Μάλτα ή στην Ελλάδα. Όμως το κλίμα εκεί είναι τέτοιο, όπου η δάσωση, εκεί όπου γίνεται, απαιτεί εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι στην Πολωνία. Τέτοιες χώρες κάνουν πολλά για να μειώσουν κατά τα άλλα τις εκπομπές τους. Άρα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα πρέπει σε θελοντική βάση να γίνεται αυτό και να επιτρέπονται διαφορετικοί τρόποι μείωσης των εκπομπών στις διάφορες χώρες. Ο κύριος Αδάσκης έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, Σαντούρσκης. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαίρετη αυτή έκθεση. Αντιλαμβάνομαι από την πλευρά μου ότι είναι πολύ χρήσιμο να έχουμε μια λογιστική καταχώρηση για τους υγρότοπους και τους βοσκοτόπους, τις εκπομπές δηλαδή από αυτούς. Και αντιλαμβάνομαι και ότι οι χώρες μέλη θα είναι οι, θα είναι οι αρμόδιες για την λογιστική αυτή καταχώρηση και όχι οι αγρότες. Αυτό μας είπε και ο Κρήτονα σήμερα. Το θέμα λοιπόν τελικά που τίθεται είναι οι αρχές πώς θα πάρουν στα χέρια τους αυτά τα στοιχεία. Εννοείται από τους ε, αγρότες. Και αυτό σημαίνει επιπλέον φόρτο εργασίας και γραφειοκρατία. Εντάξει, μεγάλες εκμεταλλεύσεις έχουν συστήματα πληροφορικής βέβαια και τους είναι πιο εύκολο. Τι θα γίνει όμως με τους μικρούς αγρότες. Γι' αυτό και εγώ προτείνω στη θελοντική βάση λοιπόν να γίνεται τέτοια λογιστική καταχώρηση στα κράτη-μέλη εφόσον θέλουν να επωφεληθούν. Με δύο λόγια προτείνω το ίδιο πλαίσιο όπως και με το πρωτόκολλο του Κιώτο. Δηλαδή η λογιστική αυτή καταχώρηση για τους ευρωτόπους και τους βοσκότοπους να γίνεται σε θελοντική βάση. Κάτι άλλο τώρα. Κάποιες άλλες πληροφορίες που θα δημιουργούσαν ε, πρόβλημα είναι η επεξεργασία. Πώς θα γίνει αυτή η επεξεργασία των δεδομένων. πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε τελικά να μην δίνουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που βασικά χρειάζονται. Κοβίτς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι φιλόδοξη η στόχη του εισηγητού μας. Πολλοί από τους στόχους του ωστόσο είναι ρεαλιστικοί. Ορισμένοι όμως δεν είναι κατά τη γνώμη μας ή τουλάχιστον δεν είναι σήμερα. Και ιδίω πρέπει να μην χρησιμοποιούμε ε, δεκαδικά στους υπολογισμούς μας, δηλαδή αντί για τόνους να, να μιλούμε σε κιλά να εκφραζόμαστε σε κιλά γιατί προσπαθούμε να τα βάλουμε όλα σε μια πολύ φιλόδοξη νομοθεσία που θα σήμαινε ότι το LULUCF είναι ήδη υποχρέωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να συνταχθούν δύο έγγραφα και μάλιστα και με χρονική διάκριση μεταξύ τους και βεβαίως να λάβουμε υπόψη και τις επιπτώσεις της νομοθεσίας αυτής. Επίσης είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ποια θα είναι η πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση και να διαρωτηθούμε είναι καλό να αναπτυχθούν τα δάση και να καταλάβουν και οι γεωργικές εκτάσεις ή είναι καλύτερα να διατηρηθούν οι γεωργικές εκτάσεις για την καλλιέργεια τροφίμων. Πρώτη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να εκφράσω τη θλίψη μου για το γεγονός ότι δεν έχουμε την οδηγία για τη διατήρηση του εδάφους που υπογράφτηκε από το Συμβούλιο. Γιατί το έδαφος είναι ένα σταθερός πόρος και δεν μπορεί να ξεφύγει ο ελεγχός του από τα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Επίσης παίζει ρόλο ε, στην αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το έδαφος. Ελπίζω λοιπόν να το λάβουμε υπόψη μας σοβαρά στο μέλλον. Τώρα, τα δορυφορικά δεδομένα όπως ακούστηκε υπάρχουν. Υπάρχουν πολύ επακριβή στοιχεία. Και θα υπάρχουν ακόμα πιο ακριβή όταν το GMS e θα, έχουν, θα είναι στη διάθεσή μας. Και επομένως δεν θα είναι πρόβλημα των γεωργών να μαζέψουν τα δεδομένα και να τα δώσουν. Μπορούν να, αν θέλουν να ενημερωθούν για τα δορυφορικά στοιχεία. Από το GMS e μπορούμε να μάθουμε πώς ο διοξίδιο του άνθρακα ε, αποθηκεύεται σε ένα δάσος το οποίο είναι καλά συντηρημένο. Επίσης, πέρα από τις δορυφορικές ε, παρατηρήσεις, θα έχουμε και παρατηρήσεις ε, in situ. Δηλαδή θα έχουμε πιλότους οι οποίοι μπορούν να παίρνουν φωτογραφίες ε, εκ του σύνεγγης που συμπληρώνουν τις δορυφορικές εικόνες και μπορούμε να βλέπουμε ας πούμε τι δεν μπορεί να κάνει ο δορυφο... και να καταγράφουμε αυτά που δεν μπορεί να κάνει ο δορυφόρος. Επομένως, μην φανταστείτε ότι οι γεωργοί, ας πούμε, βαραίνονται με αυτό το καθήκον να συλλέγουν, ας πούμε, νέα δεδομένα. Δεν ισχύει αυτό. Απλώς θέλουμε να τους εμπλέξουμε, αν θέλετε, στη διαδικασία. για την διατήρηση, ας πούμε, να τους μπλέξουμε στην προσπάθεια ε, διατήρησης του περιβάλλοντος. Ο Also ich tue mich da auch schwer. Ευχαριστώ. Βεβαίω και όποιο ασχολείται με το κλίμα σοβαρά εγκύπτει και στο θέμα Λουλουσιεφ. Βέβαια δεν είναι δυνατόν και δεν είναι και αυτονόητο. Εγώ Είμαι 40 χρόνια αγρότης και την Άνοιξη θα καλέσω τον εισηγητή στο αγρόκτημά μου. Ευχαριστώ και εσείς κύριε Πρόεδρε να έρθετε και να καθίσουμε μαζί να συμπληρώσουμε όλα τα έντυπα αιτήσεων παρόλα, παρόλα τα κομπιούτερ και τα λοιπά. Θα σας πέσει το ομολύβι από το χέρι. Θα εκπλαγείτε από ποια επιβάρυνση αντιμετωπίζουν. Και ωραία, πολύ ωραία. Έχουμε και τις ε, φωτογραφίες δορυφόρων. Έχουν όμως την ιδιότητα τα δέντρα μου να ε, πάνε και έξω από τα όρια. Επομένως παίρνει φωτογραφία από πάνω το, το δορυφόρος και τα βρίσκει τα κτήματά μου μεγαλύτερα. Και άμα δεν υπάρχει εκτιματολόγιο όπως δεν υπάρχει στη χώρα σας, να δω πώς θα λύσετε το πρόβλημα. Έχω σχεδόν την τάση να πω ότι κοιτάξτε, όταν θα υπάρχουν οι δορυφορικές φωτογραφίες και οι πληροφορίες που θα έχουμε, ή θα πρέπει να κάνουμε λεπτομερείς εκθέσεις για επιδότηση ανά εκτάριο, δεν θα υπάρχει πλέον κανένα περιθώριο. Η Κομισιόν, και μιλώ για ανθρώπους οι οποίοι είναι διπλωματούχοι γεωργοί, θα μας βάλουν όλους στο CCS, το Cross Compliance και θα είναι υποχρεωτικό μέρος των επιδοτήσεων ανά εκτάριο. Και για κάποια χρόνια θα είσαστε υποχρεωμένοι να χορηγείτε τα δεδομένα αυτά. Εγώ προτιμώ να είναι δεσμευτικά, να είναι υποχρεωτικά, διότι και η δική σας χώρα τότε κύριε Σιγητά και η Ιρλανδία και η Πορτογαλία και όλες οι άλλες χώρες θα είναι υποχρεωμένες να τα κάνουν. Προτιμώ λοιπόν να υπάρχει πλήρης εναρμόνιση. Και τι θα τα κάνετε τα δεδομένα αυτά. Χτες η Γεωργή που ήταν εδώ απ' έξω στην, ε, στην ε, πλατεία, δυστυχώς ο κύριος Λόρις μιλεί πολύ μακριά από το μικρόφωνο, έχει γυρίσει σχεδόν την πλάτη του στο μικρόφωνο, δεν τον ακούμε καλά. Μου είπαν για 4-5 χιλιάδες λίτρα ήταν γαλακτό παραγωγή. Ναι, Ωραία, τότε άμα πιούνε περισσότερο γάλα οι άνθρωποι θα έχουμε και περισσότερες αγελάδες. Τι γίνεται όμως με τα δεδομένα που συλλέγεται, θα ήθελα πολύ να το ξέρω. Είναι ανοιχτά τα πράγματα αυτά και πρέπει να συζητηθούν. Εγώ δεν θα είμαι απόλυτα κλειστός, αλλά να νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι θελοντικά και δεν θα υπάρχει καμία επίπτωση στους γεωργούς, αυτό δεν είναι αληθές. Αν κάνει σωστά τη δουλειά της Κομισιόν, μετά τα ομοσπονδιακά κρατήδια να πούν μετά στους γεωργούς ότι κοίτα πάνω στο εκτάριό σου πόσες έχεις ή πόσες δεν έχεις και θα πάνε οι γεωργοί μετά στο δάσος να μετράν τα δέντρα. Μάλιστα. Μου, άρεσε πολύ αυτά, μου άρεσαν πολύ αυτά που λες και ξέχασα να κοιτάξω και το χρονόμετρο. Να γραφτεί στα πρακτικά όμως η πρόσκληση του ε, Καρχάιντ Φλόρεντς για να πάμε στο αγρόκτημά του. Η κυρία Οκονή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Κάλς μας ε, προσκάλεσε στην ε, γεωργική του εκμετάλλευση. Το σημείωσα και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα με τον Κάλ. Απόλυτα. Δεν ακούσαμε τι υπόθηκε εκτό μικροφώνου. Συμφωνώ με τον Καρλ. Θα πάω πολύ γρήγορα, έτσι. Ανάμεσα στο 90 και το 2006, 275 εκτάρια τη μέρα λόγω της ε, διάβρωσης ε, του εδάφους και άλλων ε, προβλημάτων ε, καταστρέφονται. Επομένως, καλό είναι να έχουμε καλύτερο κτηματολόγιο, να καταγράφουμε τα δεδομένα για να βοηθήσουμε και το κλίμα. Εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να κοιτάξουμε την οικονομική επίπτωση των κειμένων που υιοθετούμε. Θα πρέπει να κοιτάξουμε την επίπτωση της διοικητικής διαδικασίας που προκρίνουμε, όπως είπε και ο Κάρλ. Η Ευρώπη σήμερα έχει μια εικόνα που είναι δύσκολο να την καταπιούν οι πολίτες μας, γιατί την περιπλέκουμε, γιατί ελέγχουμε συνέχεια, γιατί νομοθετούμε συνέχεια. Και συχνά τα κείμενά μας σημαίνουν επιπλέον διαδικασίες, επιπλέον γραφειοκρατία. Εμείς λοιπόν νομοθέτες πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το θέμα, γιατί είμαστε υπεύθυνοι για την εικόνα της Ευρώπης που προσλαμβάνουν οι πολίτες μας. Πρέπει να τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα λοιπόν. Θα πρέπει να περάσουμε σε μια ε, οικονομία χωρίς διοξείδιο του άνθρακα. Το ξέρω βεβαίως. Ε, εμείς είμαστε η, Ήπειρος, η πιο αστικοποιημένη του πλανήτη. Πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, το ξέρω. Πρέπει όμως να τα κάνουμε αυτά προοδευτικά, βαθμιδών και να κάνουμε μια προσπάθεια με βάση τους κανόνες και τις διατάξεις του Ντέρμπαν. Πιο γενικά τώρα, οι ορισμοί μας, η νομοθεσία μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι συμβατή με τους διεθνείς κανόνες, με τις διεθνείς υποχρεώσεις. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. President. Ευχαριστώ. Ακούω τη συζήτηση βλέπω ότι η εθνική μας εμπειρία, ε, το background μας, επηρεάζει το πώς αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, τα πώς τα προσεγγίζουμε. Ε, είναι πολύ περίεργο για δεδομένου του τομέα για τον οποίο συζητάμε, δηλαδή τη χρήση της γης. Ε, ούτως ή άλλως η δασοκομεία και η χρήση της γης είναι τελείως διαφορετική από κράτο μέλο σε κράτο μέλος. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η δασοκομεία έχει ένα τεράστιο δυναμικό και οικονομικό και κοινωνικό. Τα δασοκομικά προϊόντα είναι πολύ σημαντικά για τη μείωση των εκπομπών που επηρεάζουν το κλίμα. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν αυτόν τον κλάδο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η γνώση για το πώς θα το κάνουμε Ε, εξα, εξαρτάται από το ποιοι είμαστε, από πού προερχόμαστε. Είναι τελείως διαφορετική από χώρα σε χώρα, από τόπο σε τόπο. Ανησυχώ πάρα πολύ πραγματικά με κάποια τμήματα του κειμένου της Κομισιόν, όπου λέει ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν σχέδια δράσης από την Κομισιόν. Θα πρέπει να κάνει επίσης ε, συστάσεις η Κομισιόν, λες και εκείνη μπορεί να αναλύσει καλύτερα ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να χρησιμοποιηθεί αυτό το τεράστιο δυναμικό σε κάθε κρατός μέλος. Δεν συμφωνώ ότι ισχύει αυτό. Δεύτερο, σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, ο Καρλ Χάινς ε, τα είπε τόσο εύγλωτα, με τόσο ωραία παραδείγματα. Μπορεί να έχουμε δεδομένα, όντω. Αλλά πρέπει να έχουμε αξιόπιστα δεδομένα, γιατί υπάρχουν και λιγότερο αξιόπιστα δεδομένα. Και υπάρχουν και δεδομένα που είναι σκουπίδια. Ε, είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα αξιόπιστα δεδομένα. Γιατί αν αρχίσουμε να τα μπλέκουμε όλα, νομίζω ότι θα κάνουμε περισσότερο κακό παρά καλό. Θα περιπλέξουμε τα πράγματα και ο αγώνας ε, για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή θα γίνει πιο δύσκολος. Το συμπέρασμά μου λοιπόν είναι να μην κάνουμε τον Τέρμπαν ε, Λουλουσιέφ ε, να το κάνουμε να δημιουργήσει δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δηλαδή κανόνες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και κανόνες για τους υπόλοιπους. Ο Πίτερ Λίζε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καθώς και όλους τους συναδέλφους για την ζωηρή συζήτηση. Συμφωνώ με εκείνους που είπαν ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λέει η Κομισιόν ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση για τους αγρότες, δεν μου αρκεί αυτό. Γι' αυτό και μαζί με τον εισηγητή έχω καταθέσει την τροπολογία 79 και θα παρακαλέσω για υποστήριξη από όλους τους συναδέλφους και θέλω να ακούσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν μπορεί να αποδεχτεί την τροπολογία αυτή, διότι τότε θα έχουμε μεγαλύτερη σαφήνεια. Γιατί όποιο Γιώργο θεωρήσει ότι είναι σημαντική επιβάρυνση που του επιβάλλουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να επικαλεστεί αυτή την ε, τροπολογία. Να ε, προσέξουμε επίσης τα όσα είπαν και προηγουμένω άλλοι συνάδελφοι για το διπλό, διπλή καταμέτρηση. Έχουμε και τη βιομάζα και ίσως πρέπει να αλλάξουμε κάτι και στο, ευρωπαϊκό, και στο, ε, σύστημα ε, εμπορίας ε, εκπομπών. Τώρα, μακροπρόθεσμη στόχη δεν μπορεί παρά να είναι οι αγρότες και οι δασοκόμοι που παίζουν πολύ θετικό ρόλο στην προσπάθεια αντιμετώπισης αλλαγής του κλίματος να ε, αναγνωριστεί ο ρόλος αυτός. Επαναλαμβάνω ότι οι αγρότες ήδη συμβάλλουν σημαντικά στην διατήρηση του κλίματος και αν τους ενισχύσουμε περισσότερο εφόσον ανταποκρίνονται καλύτερα στα καθήκοντά τους, τόσο το καλύτερο. Έρχομαι σε αυτά που είπε η κυρία Κλάς και θα παρακαλέσω να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από όσο γνωρίζω, ένα βιώσιμα καλλιεργούμενο δάσος αποδίδει περισσότερο από ένα δάσος το οποίο αφήνεται να αγρέψει. Όχι λοιπόν μονάχα ζούγκλα και φυσικά πάρκα, αλλά και το καλά ε, διατηρημένο δάσος. Αυτό να περιληφθεί και στις προτάσεις του κ. Τσιόλος. Αυτά που λέμε εμείς αλλά και η Επιτροπή Γεωργίας για να έχουμε τελικά μια συνολική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στους Γεωργούς. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Κομισιόν που εκπροσωπείται σήμερα τον κύριο Όλσεν. Σας παρακαλώ όχι πάνω από τρία λεπτά. Έχουμε μια ακόμα σημαντική έκθεση σήμερα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, για την τόσο ζωντανή συζήτηση που είχαμε μέχρι τώρα και για τις πολλές τροπολογίες. Πολλές από αυτές είναι πάρα πολύ χρήσιμες γιατί αποσαφηνίζουν το κείμενο και προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας όλες σας τις ανησυχίες. Τώρα θέλω να είμαι ευθύ μαζί σας όσον αφορά το άχθος που επομίζονται οι αγρότες. Ναι, μπορούμε να δεχτούμε την τροπολογία την 79. Και εγώ έρχομαι από μια οικογένεια αγροτών στη Δανία. Η Δανία κάνει αυτή τη λογιστική καταχώρηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τον ρωτάω τους αγρότες στην οικογένειά μου αν το ξέρουν ότι γίνεται αυτό, δεν το ξέρουν. Αν τους ρωτάω αν οι ίδιοι συμπληρώνουν τίποτα έντυπα γι' αυτό, λένε όχι. Αν ε, απευθυνθείτε στην Ένωση των Αγροτών, Κανένας δεν έχει πάει να τους μιλήσει, κανένας αγρότης δεν έχει παραπονηθεί για αυτή τη λογιστική καταχώρηση. Όλα αυτά τα στοιχεία λοιπόν συλλέγονται μέσω άλλων καναλιών, μέσω άλλων συστημάτων συλλογής δεδομένων, είτε μέσω της κοινωνικής πολιτικής, είτε μέσω της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Και είναι κάτι υποχρεωτικό εδώ και 20 χρόνια τα κράτη-μέλη ήδη κάποια από αυτά τα δεδομένα τα δίνουν ήδη. Και απλώς συμπληρώνονται από άλλες πηγές τώρα. Δηλαδή με δύο λόγια πρέπει να πούμε ότι δεν θα υπάρξει επιπλέον άγχος από αυτήν εδώ τη ρύθμιση. Βέβαια το δεύτερο στάδιο, όταν θα συζητήσουμε στόχους, τότε θα γίνει παρετέρω η συζήτηση και τότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Κατόπιν τούτον, για τις τροπολογίες, θέλω να σας πω γενικά ότι, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι τεχνικό το ζήτημα. Και γι' αυτό το θέμα πρέπει να μείνουμε στα πλαίσια της απόφασης που είχαμε την προηγούμενη χρονιά στον Τέρμπαν. Πολλές από τις τροπολογίες λοιπόν προσπαθούν να προσεγγίσουν το κείμενο στον Τέρμπαν. Για κάποιες άλλες θα πρέπει να σας πω ότι εμείς η Επιτροπή υποψιαζόμαστε ότι δεν θα είναι παραδεκτές. Αυτό φοβόμαστε. Δυστυχώς για τα προϊόντα δασοκομείας πρέπει να σας πω ξυλίας, υλοτομία οι 235 και 236 και οι 223 είναι σε αντίθεση με το διεθνές πλαίσιο το οποίο έχουμε ήδη συνυπογράψει. Οπότε σας παρακαλώ να τις ξανασκεφτείτε. 233. Δεν είναι σε αντίφαση μεν, αλλά μας κάνει να δημιουργούσε επιπλέον ε, καταχώρηση και επιπλέον ε, δυσκολίες για τα προϊόντα ελοτομίας. Προσπαθώ να σας μεταφέρω ένα σαφές μήνυμα. Να υπογραμμίσω ότι δεν λέω πολιτικά, δεν κάνω καμία πολιτική κρίση, απλώς σας λέω ότι πρέπει να ευθυγραμμιζόμαστε με τις διεθνείς συμφωνίες. Και τέλος, η λογιστική καταχώρηση από τις ε, γεωργικές δραστηριότητες. Αυτό είναι κάτι που άλλες χώρες το κάνουν, άλλες όλοι. Πολλές χώρες δίνουν πάρα πολλά δεδομένα ήδη και το κάνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό και τα δίνουν στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Συνεπώς, το θέμα δεν είναι αν υπάρχουν ε, τα στοιχεία ή δεν υπάρχουν, είναι πολιτικό το ζήτημα το οποίο καλείστε να αποφασίσετε. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Τώρα. Um, Μια συγκεκριμένη ερώτηση υπήρξε και από την κυρία Κλάς και από μένα. Μπορείτε να την απαντήσετε παρακαλώ. Ο πρόεδρος, μήπως γίνεται διμερός μετά, γιατί θα ήθελα να δώσω το λόγο στον εισηγητή πρώτα. Ο εισηγητής. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για το ενδιαφέρον που δείχνουν για το θέμα μας. Δεν θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση τους μύθους και τους φόβους μας. Κάνουμε Ούτω ή άλλω αυτή η προσπάθεια λογιστική καταχώρηση είναι κάτι που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία κράτη-μέλη το κάνουν ήδη. Α πούμε η Δανία είναι μία από αυτέ τι χώρε. Και δεν βάρινε σε καμία περίπτωση του ε, γεωργού. Οι διοκτήτες δασών είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αυτή τη λογιστική καταχώρηση. Ούτως ή άλλω δεν μιλάμε για αυτούς. Μιλάμε για την ε, υποχρέωση που θα βαρύνει του γεωργού για την λογιστική καταχώρηση ε, των γεωργών. Για τους ιδιοκτήτε δασών δεν αλλάζει τίποτα. Ήδη γίνεται αυτό, επαναλαμβάνω. Τώρα, ποιο είναι το διακύβευμα. Το αν θα καταδείξουμε, αν θα φανούν οι οικονομίες που κάνουμε. Γιατί αν το κάνουμε θα έχουμε σαφές οικονομικό πλεονέκτημα. Και αυτό το πλεονέκτημα περνάει στα κράτη-μέλη. Είναι προ όφελο των κρατών μελών. Κυρία Χιούμπνερ, για τα πολωνικά δεδομένα. Σα ευχαριστώ καταρχά για τα σχόλιά σα. Η Πολωνία από τις ετήσιες εκπομπές της θα γλιτώσει το 1% θα κερδίσει το 1%. Αυτή τη στιγμή καταχωρήσετε και αυτές τις ε, εξοικονομίες. Και η Σουηδία. Η Ιταλία θα γλιτώσει 2% από τις βιομηχανικές εκπομπές. Χάρη ε, στην προσπάθεια της ε, Σιέφ. Αυτό σημαίνει και λεφτά πέρα από όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, θα πρέπει να βοηθήσετε τις ε, χώρες. Αν θέλετε να βοηθήσετε τις χώρες σας και τον λαό σας, θέλω να σας πω ότι κανένας αυτή τη στιγμή στο γεωργικό τομέα δεν πιστεύει ότι θα υπάρξει γραφειοκρατία λόγω αυτού. Αρχικά πίστευε κάτι τέτοιο ο γεωργικό κλάδο. Το πίστευε πριν από τρει μήνε. Αλλά όποιο ε, κάνει μια συζήτηση τώρα με του γεωργού θα προκύψει ξεκάθαρα ότι δεν εισφίσταται αυτό. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα γραφειοκρατίας. Ε, το θέμα είναι αυτή την εξοικονόμηση που κάνουμε ούτω ή άλλω λόγω του Λουλουσιεφ. Θα την αφήσουμε να παραμένει κρυφή και αόρατη. Δεν θέλουμε να την ε, ε μετρήσουμε και αυτή. Δεν θέλουμε να την υπολογίσουμε. Ευχαριστώ, Κρήτονα. Σε ευχαριστώ για αυτά τα συμπεράσματα που βγάζει για τη συζήτηση. Στις 10 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή ΕΜΒΗ. Και τον Ιανουάριο του 2013, κανονικά, θα πάει το σημείο αυτό στην Ολομέλεια. Κανονικά, έτσι. Ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Και συνεχίζουμε τώρα. Έκθεση Περέλο για το θόρυβο στα αεροδρόμια. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό θα προσπαθήσω να συνοψίσω όσο μπορώ πιο σύντομα για να μπορέσουν όλοι να αντιδράσουν. Λοιπόν, όπως όλοι γνωρίζετε, για την στην έκθεση βεβλήθησαν 80 τροπολογίες. Οι περισσότερες από αυτές πρέπει να σας πω ότι μπορούμε να τις δεχτούμε. Και οι περισσότερες βελτιώνουν ακόμα περισσότερο το κείμενο. Είναι μεγάλος βέβαια αριθμό των τροπολογιών, αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι πολλές από αυτές ε, καταδίδεται σε εντελώς διαφορετικά άρθρα. Πράγμα το οποίο μας δυσκολεύει κάπως, γιατί ναι, μερικέ είναι για το άρθρο 5, άλλε όμως ε, μας δυσκολεύουν να καταλήξουμε σε συμβαστικέ τροπολογίες γιατί δεν μπορούμε να συγκεντρώσουμε τις τροπολογίες αφού πάνε προ πάσα κατεύθυνση. Στο άρθρο 4 σημείο 5 για παράδειγμα και κάποια άλλη υπάρχει μια προφορική που μας δυσκολεύει. Κατά τα άλλα, όπως σας είπα, μπορούμε να τις δεχτούμε ως έχουν. Όμως, όμως, Νομίζω παρόλα αυτά ότι θα έπρεπε να ξαναδούμε κάπως τις τροπολογίες επί του κειμένου της Επιτροπής της δικές μου. Κυρίως εκεί που ενδιαφερόμαστε, ε, στα, που ασχολούμαστε με τα διαφερόμενα μέρη, την επανεισηγωγή δηλαδή του ορισμού των διαφερόμενων μερών. Στο άρθρο 5 και στο 7 θα δείτε ότι τονίζουμε το σημείο αυτό των ενδιαφερομένων μερών. Και στο άρθρο 10 με σαφήνη ορίζουμε το δικαίωμα των ενδιαφερόμενων μερών να ελέγχουν τις δραστηριότητες από την ηχορύπανση των αεροσκαφών. Εμείς ε, προτείνουμε κάποιες τροποποίησεις στο κείμενο, στο κείμενο λοιπόν της Επιτροπής ο έλεγχο να μην είναι αποκλειστικά στην Επιτροπή, αλλά να υπάρχει δυνατότητα να εξετάζουν και τα διαφερόμενα μέρη και να προτείνουν αλλαγέ. Το κείμενο τη επιτροπή έχει αυτό το άρθρο λοιπόν και τι ε, προτάσει για κατάργηση των διαφερόμενων μωρών, ενώ το δικό μα κείμενο πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλά ισορροπημένο. Σκεφτόμαστε το θέμα αυτό της κατάργησης και πιστεύουμε ότι θα δημιουργούσε ένα κενό το οποίο θα είχε αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που θεωρητικά θέλουμε να πετύχουμε με την ε, πρόταση αυτή. Τώρα υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που θα έπρεπε να τις δούμε και από νομική άποψη. Έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας απαντήσει γι' αυτά. Έχω σας λέω αμφιβολίες για την νομική πτυχή. Ακόμα και αν πολιτικά συμφωνώ μαζί τους. Το θέμα της χωροταξίας, για παράδειγμα. 66, 67, 84, 71 της κυρίας Γιανακουδάκη που προτείνει μια τροποποίηση στα επίπεδα δεσιμπέλ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να το δεχτούμε αυτό σε μια τέτοια πρόταση τη στιγμή που τροποποιείται η αρχική για την ε, ηχορύπανση οδηγία. Πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι συμπληρωματική η πρόταση αυτή και συγκεκριμένα για την ε, αεροπλοία μια που προσπαθεί να ελέγξει την ηχορύπανση. Να μην μπερδεύουμε δηλαδή τα μέτρα που προτείνουμε για την τροποποίηση των κριτηρίων ηχορύπανσης έτσι όπως υπάρχει σε άλλη οδηγία. Όταν εμείς μιλήσαμε για την ε, δημόσια συμμετοχή ή των ενδιαφερόμενων μερών ήταν πιο πολύ για να υπάρχει μια συμμετοχή και έτσι να ακούγεται και άποψη όλων των πλευρών και να υπάρχει διαφάνεια. Γι' αυτό και θέλω να διακρίνουμε τα δύο πράγματα, γιατί δεν μπορεί να ζητάμε μια τεχνική άποψη από τον εκπρόσωπο κάποιου ενδιαφερόμενου μέρους που μπορεί να μην γνωρίζει αυτά τα τεχνικά στοιχεία. Είναι κάτι διαφορετικό αυτό. Κάτι άλλο που πρέπει να σκεφτούμε είναι τα παραρτήματα 1 και 2. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, εγώ πρότεινα να διαγραφούν τα παραρτήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση της χορύπανσης και τη σχετική οδηγία. Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ περιοριστικό, γιατί σας είπα ότι δεν τροποποιούμε την οδηγία αυτή. Ούτε έχουμε δύο σε εθελοντική βάση οδηγία ή τη μία ή την άλλη. Όχι, και οι δύο είναι υποχρεωτικές. Η μία συμπληρώνει την άλλη. Τα παραρτήματα διευκρινίζουν ότι δεν μιλάμε γενικά για την ηχορύπανση, αλλά για την ηχορύπανση που προκαλείται από τα αεροσκάφη. Γι' αυτό και σας ζητάω να το σκεφτείτε, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο μας με τα παραρτήματα αυτά. Επίσης θέλω να σας πω ότι οι προτάσεις μου φαίνονται σωστές. Βέβαια για τη γνωμοδότηση έχω δουλέψει πολύ. 80 τροπολογίες μπορεί να σας φαίνονται πολλές και είναι πολλές για μια γνωμοδότηση πράγματι. Πάντως τόσο οι σκιώδες εισηγητές όσο και οι συνάδελφοι που έκαναν τον κόπο να υποβάλουν τροπολογίες να ξέρετε ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά και θέλω όλους αυτούς να τους ευχαριστήσω και να τους πω ότι συμφωνώ μαζί τους. Θα τους στείλω τις ε, προσπάθειες που μπορώ να κάνω για συμβαστικές τροπολογίες και ποιες πιστεύω ότι πρέπει να παραμείνουν για τη βελτιώνει το κείμενο. Αυτά για την γνωμοδότησή μου. Και επίσης θα σας πω και ποιες θεωρώ παραδεκτές και ποιες όχι. Θα σας τα στείλω όλα αυτά για να κερδίσουμε χρόνο τώρα και να μην σας πω πολύ περισσότερο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλώς. Μπαίνουμε τώρα στη συζήτηση. Η κυρία Κλάς πρώτη. Ευχαριστώ καθώς και τον εισηγητή. Και βεβαίως και για τη θετική του στάση απέναντι στις τροπολογίες. Και το επιστρέφω τη φιλοφρόνηση διότι είναι και καλή η πρόταση του εισηγητού. Μένει ανοιχτό το ερώτημα, αν θέλουμε κανονισμό ή οδηγία. Εγώ τάσομαι υπέρ του κανονισμού, διότι επιτρέπει ευθύτερη, αμεσότερη εφαρμογή. Ο θόρυβος έχει μεγάλο ενδιαφέρον και κοινωνικό. Θα δείτε και από τα ηλεκτρονικά ταχυδρομεία που λαμβάνουμε, που είναι ιδιαίτερα έντονα και ρωτούν «Μα πώς γνωμοδότηση μόνο της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Προστασίας της Υγείας» διότι θεωρούν ότι ο θόρυβος είναι ιδιαίτερη επιβάρυνση. Διότι μπορεί μεν να μετρά κανείς το θόρυβο αντικειμενικά με μετρήσεις, αλλά η υποκειμενική πρόσληψη της ενόχλησης είναι κάτι το οποίο ξεφεύγει από τις μετρήσεις. Και οι ενδιαφερόμενοι θέλουν, ζητούν να τους ακούσουμε. Εγώ είμαι βέβαια ότι η απέτηση όλων των ενδιαφερομένων είναι να μειωθεί ο θόρυβος. Και το επιζητούν αυτό και οι αεροπορικές εταιρείε και οι φορείς των αεροδρομίων. Δηλαδή η αποδοχή είναι γενική. Πολλές τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Εγώ παρετήρησα ότι υπάρχουν και πολλές τροπολογίες οι οποίες στρέφονται κυρίως γύρω από την αποδοτικότητα των ε, ε, μέτρων θα πρέπει να μιλούμε για τα, για, τις, για τα αποδοτικότερα μέτρα και οικονομικά αλλά και από τις άλλες απόψεις, από την απόψη της αποτελεσματικότητας. Εγώ προτείνω, και το είπε και ο εισηγητής, να παραπέμψουμε ευθέως στην οδηγία του 2002 για τον θόρυβο από πηγές του περιβάλλοντος διότι είναι σαφές ότι εδώ προέχει η προστασία της υγείας. Και εκεί προβλέπεται διαφανής διαδικασία με συμμετοχή των πολιτών. Και αυτό επιζητούμε και εδώ. Και οι αρμόδιες αρχές των χωρών μελών καλούνται να κάνουν τακτικά τον σχεδιασμό, να καταθέτουν σχέδια δηλαδή προστασίας κατά του θορύβου. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία περιλαμβάνουμε και εμείς και συζητούμε και στην οδηγία αυτή. Τα παραρτήματα 1 και 2 του σχεδίου κανονισμού προβλέπουν και σχέδια δράσεως της οδηγίας για τη μείωση του θορύβου. Έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την δαπανηρή επικάλυψη των νομοθετημάτων και να βελτιώσουμε την ε, προστασία από τον θόρυβο. Αυτό είναι νομίζω που ενδιαφέρει και στην οδηγία προστασίας από τον θόρυβο του περιβάλλοντος λέει καθαρά ότι η διασφάλιση υψηλού επίπεδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος αποτελεί τμήμα της κοινοτικής πολιτικής και ένας από τους στόχους είναι και η προστασία από τον θόρυβο. Ο στόχος είναι λοιπόν η κοινή ανάπτυξη ε, σχεδίων για την απάλυνση ή για την μείωση του θορύβου. Πρόκειται δηλαδή για ε, διατάξεις οι οποίες είναι θετικές και οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως βάση. Είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν τα αιτήματα των τοπικών αρχών που είναι βεβαίως στην καλύτερη κατάσταση να γνωρίζουν ε, το τι συμβαίνει στα αεροδρόμια της περιοχής τους. Οι επιδράσεις είναι άλλωστε τοπικού χαρακτήρα και γι' αυτό πρέπει οι σχετικές αποφάσεις να ληφθούν επιτόπου και με συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού. Να προβλέψουμε δηλαδή συγκεκριμένε λύσεις για τα προβλήματα επιτόπου και αυτές να εγκριθούν. Υπάρχει και μέγα κύμα των αντιτιθέμενων που λένε ότι δεν μπορεί η Κομισιόν να, είναι το τελευταίο, να έχει τον τελευταίο λόγο διότι τότε αυτό ακυρώνει όλα τα ε, ενδιάμεσα βήματα τα οποία κάνουμε εμείς δηλαδή διαμεσολαβούμε μεταξύ των αρχών του κοινού κτλ. εμείς ως ευρωβουλευτές και τελικά αν η Κομισιόν έχει τον τελευταίο λόγο και έλθει και τα απορρίψει ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν να το προσέξουμε. Επίσης οι αεροπορικές μεταφορές έχουν και περιφερειακό χαρακτήρα αλλά και καθαρά υπερπεριφερειακό χαρακτήρα. Η μείωση του θορύβου των αεροσκαφών επίσης πρέπει να προωθηθεί. Είναι βέβαια μακρόχρονη διαδικασία διότι πρέπει να γίνουν προμήθειες νέων αεροσκαφών και να παροπλιστούν τα παλαιά. Επίσης υπερπεριφερειακά πρέπει να γίνουν τα σχέδια των, ε, ε, να σχεδιαστούν δηλαδή οι αεροδιάδρομοι που κινούνται τα αεροσκάφη. Όταν το αεροσκάφος απογειώνεται πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά και ποια ε, διαδρομή θα ακολουθήσει και πού θα καταλήξει να προσγειωθεί. Το ίδιο πρέπει και να προβληθούν ε, χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι. Βεβαίως και πάση συζητηθούν αυτά και με τις ε, ε, αεροπορικές εταιρείες. πρέπει να γίνει συντονισμός μεταξύ των περιφερειών. Δηλαδή, οι συνθήκες από και προς πρέπει επίσης να είναι απολύτως ξεκάθαρες. Χρειάζεται και ρύθμιση για την οικονομική, πέραν μάλλον από την οικονομική αντιμετώπιση των ε, αεροπορικών εταιριών. Χρειάζεται συντονισμός μεταξύ τους. Γνωρίζω ότι από πλευρά των αεροπορικών εταιριών έχει προωθηθεί η υπόθεση αυτή, αλλά χρειαζόμαστε βεβαίω περισσότερα βήματα να γίνουν για να υπάρξει μεγαλύτερο συντονισμό και έτσι να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σύνολο δράσεων στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίω. Κοιτάζω λίγο το ρολόι, λέει ο Πρόεδρο, διότι ε, δεν θα προλάβουμε. Chris Davis που ε, εκπροσωπεί άλλη σκιώδη ιδρία. Εκπροσωπώ την, ε, τον Ανδρέα Ζανόνη. Θέλω να πω στην Επιτροπή ότι ο κύριος Ζανόνη μου είπε ότι είναι μια γνωμοδότηση, έχουμε ευθύνε για την υγεία και η βασική εστίαση δική μας θα πρέπει να είναι στην υγεία των πολιτών και πώς μπορεί να επηρεαστεί από τον θόρυβο των αεροδρομίων. Επηρεάζεται ήδη από την μόλυνση της ατμόσφαιρας και από τη χημική μόλυνση. Γενικά είναι υπέρ της προσέγγισης του εισηγητή με τις τροπολογίες του θέλει να συμπληρώσει αυτή την ε, νομοδότηση. Και η μελέτη αντικτύπου στο περιβάλλον ε, και μέτρα μείωση του θορύβου ε, θα πρέπει να γίνεται με συστηματικό τρόπο. Ε, η ενεργή συμμετοχή των πολιτών να υποστηρίζεται από όλε τι πολιτικέ ομάδε. Χαίρεται γι' αυτό. Η αξιολόγηση του θορύβου και η συλλογή των δεδομένων θα πρέπει να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια. Συμφωνεί με αυτό. Αλλά το βασικό θέμα τη τροπολογία 1 είναι αν θα πρέπει να έχουμε εδώ κανονισμό ή οδηγία. Διαφωνεί με τον εισηγητή και πιστεύει ότι η Κομισιόν ορθά προτείνει κανονισμό γιατί είναι το πιο αξιόπιστο και εναρμονισμένο εργαλείο και η νομική βάση που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε. Α, τώρα να σας μιλήσω και με τις, για τις δικές μου απόψεις. Συμφωνώ με τον κύριο Σανώνη ότι όντω αυτό είναι ένα αρμονισμένο και αξιόπιστο νομικό πλαίσιο, φαντάζομαι ότι και στη δική μου ομάδα για λόγου ε, επικουρικότητα και αναλογικότητα μπορεί να αμφισβητηθεί λιγάκι αυτό, αλλά εγώ πάντω έχω αυτή την άποψη. Ότι είναι καλύτερο ο κανονισμό. Ευχαριστώ. Τον Κρι. Ποιο είναι ο επόμενο ομιλητή, η κυρία Γιανακουδάκη. Οι πράσινοι λείπουν, ε. Εγώ θέλω να μιλήσω για το περιβάλλον. Μόνο. Συμφωνώ με τον Κρίς μάλιστα, με τους συμμάχους μας. Θα πρέπει να δούμε το θέμα από τη σκοπιά της υγείας των πολιτών. Ε, το περιβάλλον, η βιομηχανία και οι πολίτες είναι τρεις τομείς που προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Ε, φυσικά ε, δεν υπάρχει μαγική λύση για όλα. Ένα από τους τομείς που θέλουμε διευκρινήσεις και θα υποβάλουμε τροπολογίες είναι ο ορισμός των διαφερομένων μερών. Και ποιος μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Ποιοι είναι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι. Με την τροπολογία μας νομίζω το ρυθμίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό το σημείο και ελπίζω να την υποστηρίξετε. Θα σταματήσω εδώ για να αφήσω και άλλους να μιλήσουν. Äh, Ευχαριστώ. Εκατοντάδες email λαμβάνουμε από πολίτες που ανησυχούν και ε, που ζητούν βελτίωση της προτάσεως. Ανησυχούν για το ότι παίρνει δευτερεύουσα θέση η προστασία της ε, υγείας και ότι κυρίως μας απασχολούν τα στοιχεία κόστους. Κατανοώ, άλλωστε και εγώ κατοικώ κοντά σε αεροδρόμιο, κατανοώ λοιπόν τις ανησυχίες τους. Πάντοτε είπα ότι ε, η ποιότητα ζωής και η υγεία πρέπει να είναι υπέρτερη στόχη από το κέρδος. Δεν αρκούν οι προτάσει της Κομισιόν για τη μείωση του θορύβου. Δυστυχώς η βελτίωση της προστασίας θορύβου παίζει δευτερεύοντα ρόλο στην πρόταση της Κομισιόν. Αυτό που ενδιαφέρει την Κομισιόν είναι καθαρό στο εκτιμώντας εννέα. Τα μέτρα μείωση του θορύβου θα πρέπει να μπορούν να ε, αναστέλλονται εφόσον βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων. Υπάρχει σχετική τροπολογία που βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση αλλά όχι επαρκώς. Γι' αυτό εγώ θα ζητήσω να διαγραφεί το εκτιμώντας αυτό όπως ζητεί ο εισηγητής. Επίσης χαιρετίζω την πρόταση του ε, εισηγητού για μέτρα μείωσης του θορύβου με διακοπή λειτουργίας ε, ορισμένων ε, διαδρόμων προς και απογειώσεως. Νομίζω ότι η προστασία της υγείας και της ευημερίας των πολιτών πρέπει να μας απασχολούν πρωτίστως. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι ουσιαστική σημασία να συμμετάσχουν και οι φορείς των αεροδρομίων, να τους ακούσουμε. Ο στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι αυτός. Θεωρώ ότι είναι αμφίβολο εάν αυτός αυτή η πρόταση κανονισμού που κυρίως ε, ασχολείται με την μείωση του κόστους μπορεί να θεωρηθεί ισορροπημένος. Και γι' αυτό προτείνω εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας. Επίσης, ζητώ ότι το άρθρο 4 παράγραφος 2 πρέπει να διαγραφεί. Η πράξη έδειξε ότι μείωση λειτουργίας πρέπει αντίθετα με το προτινόμενο αυτό κείμενο πρέπει να είναι από τα πρώτιστα μέτρα. Εν τέλει, δύο ακόμα θέματα. Θεωρώ ότι με τη μείωση λειτουργίας στη βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων πρέπει με αυτόν τον τρόπο να λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και γι' αυτό το άρθρο 10 για την αρμοδιότητα ελέγχου θεωρώ ότι είναι περιττό. Το ίδιο για την προστασία των ε, δικαιωμάτων των χωρών μελών θεωρώ ότι πρέπει να διαγραφούν τα σχετικά με την υποχρεωτική ανακοίνωση. Ε, στην κοινοποίηση μάλλον στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο εσείς κυρία μου, αλλά πολύ σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή για όλα όσα μας είπε. Συμφωνώ απόλυτα με πολλούς από τους ομιλητές που λένε ότι πρέπει να πρόκειται για οδηγία. Όντως εδώ τίθεται ένα μεγάλο θέμα αρχής επικουρικότητας, οπότε ναι, πιστεύω και εγώ ότι πρέπει να παραμείνει οδηγία. Τώρα για τα διαφερόμενα μέρη που αναφέρθηκαν. Ποια πρέπει να είναι τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για μένα θα πρέπει να είναι εκλεγμένοι από δημοτικά συμβούλια για παράδειγμα και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ποιους θα βάζουμε μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Τώρα, η δυσκολία με το θέμα του όρου υγεία είναι ότι ποσοτικά είναι δύσκολο να εκφραστεί. πρέπει να έχουμε υπόψη μας τα μέτρα για την κυκλοφορία των ορασκοφών, την υποδομή και όλα αυτά πράγματα, τα οποία εννοείται ότι επηρεάζουν τον βαθμό της συγχωρήπανσης και άρα τις επιπτώσεις στην υγεία. Επίτα νομίζω ότι μόνο για τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να μιλάμε εδώ. Τώρα ο λέει και κάτι άλλο πολύ καλό. Ε, αναφέρθηκε στα decibel, το επίπεδο των δεσιμπέλ. πόσο, 10, 15, τι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας να πούμε ποιο είναι το σωστό νούμερο. Πρέπει να δούμε τι υπάρχει στη θέση μας μέχρι τώρα. Τέλος, Πρόεδρε, μην ξεχνάμε ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια αποτελούν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο των υποδομών μας. Υπάρχουν ε, μεγάλες, μικρές εταιρείες, πολύ συχνά μικρές, παλιά αεροσκάφη πολλές φορές. Βοηθούν όμως από την άλλη μεριά τον κόσμο να μετακινείται. Ο κλάδος θέλει μια ισορροπημένη προσέγγιση. Θέλει σωστέ προδιαγραφέ. Οι συζητήσει που γίνονται στο Συμβούλιο μέχρι τώρα, πόσο ξέρω, πηγαίνουν προ τη σωστή κατεύθυνση. Συνεπώ, για άλλη μια φορά, ευχαριστώ τον εισηγητή. Σίγουρα κάποιοι θα συμφωνήσουν ή θα διαφωνήσουν με το ένα ή το άλλο σημείο, αλλά τελικά και γενικά νομίζω ότι πρέπει να πούμε ότι και στην Επιτροπή Μεταφορών είχαμε πολύ καλή συζήτηση για το θέμα αυτό και έτσι πιστεύω να καταλήξουμε θετικά. Εδώ εξαντλήθηκε ο κατάλογος των αγορητών για τις απαγορεύσεις νυχτερινών πτήσεων. Διότι βεβαίως όταν ε, επιβάλλεται μια απαγόρευση νεκτερινών πτήσεων τότε μεταφέρονται οι νεκτερινές πτήσεις σε άλλα ε, σε άλλα ε, τμήματα, του, σε, άλλα μέρη. Ε, θα δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, που είναι ο, ο Διευθυντής από τη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών. Ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία στην Επιτροπή να σχολιάσει. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον ε, κύριο Περέγιο Ροντρίγκης αλλά και τους σκιώδες εισηγητές για τη δουλειά που έκαναν σε βάθος. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί τα έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Από αυτά που είπατε. Αυτό που με κάνει να αντιδράσω κυρίω είναι το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής. Θέλω να σας πω ότι η Επιτροπή συμμερίζεται απόλυτα την ανησυχία σας. Αυτή και για την Επιτροπή, είτε και για οποιαδήποτε αρχή, είτε ευρωπαϊκή, είτε περιφερειακή. Αυτό είναι το βασικό πράγματι. Οπότε η πρόταση αυτή, αυτό το νομικό μέσο, η πρόταση που έχουμε, στην οποία έχουμε καταλήξει, πώς θα λάβει καλύτερα υπόψη τις ανησυχίες αυτές για την υγεία. Η πρότασή μας αναφέρεται στην αεροπλοία και στην διαδικασία που θέλουμε να ακολουθήσουμε άπαξ οι εθνικές οι περιφερειακές αρχές αποφασίζουν για ε, περιορισμούς. Η πρότασή μας δηλαδή προσπαθεί να συνδέσει τα διάφορα επίπεδα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, το τοπικό, το εθνικό, το ευρωπαϊκό και όπου και το διεθνές. Πώς λοιπόν αυτές τις ανησυχίες για την υγεία και την ασφάλεια μπορούμε να τις συμπεριλάβουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία, τηρώντας τις ε, διαδικασίες το δίλημα, υπάρχει λοιπόν το δίλημα που λέει ότι θέλουμε να κάνουμε πιο αυστηρέ τι προδιαγραφέ και από την άλλη μεριά να τηρούμε την οδηγία για την ηχορύπανση. Ακούσαμε τον εισηγητή που λέει ότι πρέπει να είναι συμπληρωματικά αυτά τα δύο μέσα. Η οδηγία λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να εντοπίζουν τις πηγές συγχωρήπανσης, να χαρτογραφούν την κατάσταση, να υιοθετούν προγράμματα δράσης για να καταπολεμήσουν την ηχορύπανση βάση τεχνικών μετρήσεων η χορύπανση. Τώρα, το, εμείς το λέμε κάπως διαφορετικά. Θέλουμε να είναι ένα toolbox για να εφαρμόζονται οι μετρήσεις αυτές και που να συμμορφώνονται βέβαια με τις διεθνείς προδιαγραφές εννοείται. Εμείς δεν προσπαθούμε να το αφαιρέσουμε αυτό που λέτε εσείς για τα κράτη-μέλη, ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να θέτουν στόχους που μπορεί να έχουν και άλλους που είναι η περιφερειακή τους ανάπτυξη, αλλά επιπλέον προτείνουμε μία διαδικασία για τα διάφορα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, για το κόστος τους, για την αποτελεσματικότητά τους τι συνδυασμό μέτρων ενδεχομένω θα μπορούσε να υιοθετήσει κάποιο κλπ. Δηλαδή για να είμαστε ξεκάθαροι, Εμεί πιστεύουμε ότι το ευρωπαϊκό περιβάλλον για την ηχορύπανση, πλαίσιο μάλλον πιο σωστά, είναι το καταλληλότερο. Και θέλουμε να λαμβάνεται υπόψη και η σχέση ε, κόστους και αποτελέσματος. Γιατί το κόστος είναι σημαντικό, όντως. Από την άλλη είναι δύσκολο, όπως είπε και κάποιος, να εκφράσουμε ποσοτικά την υγεία. Γίνεται λοιπόν μια σύνδεση ανάμεσα στην ηχορύπανση και το περιβάλλον. Τώρα, ναι, θα είμαι σύντομος. Δύο άλλα πραγματάκια τα οποία ακούσαμε εδώ σήμερα. Το πρώτο έχει να κάνει... Έχει να κάνει με τη συμμόρφωση των ε, αεροσκαφών. Τι περιθώριο υπάρχει είναι γεγονός ότι τα πιο μεγάλα, τα πιο χειρά αεροπλάνα είναι αυτά που προκαλούν και τη μεγαλύτερη ηχορύπανση. Θέλουμε εμείς να εισαγάγουμε έναν ορισμό για τις εθνικές τοπικές αρχές, ώστε όταν εξετάζουν τους περιορισμούς για την ηχορύπανση, να έχουν αυτόν τον ορισμό που θα κάνει τη διαφορά για τις επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια. Μπορεί να υπάρχει κάποια σύγχυση εδώ. Πάντω οι τροπολογίε που προτείνονται, που μιλάνε για το μείον 8 ή μείον 10, αυτό αφαιρεί από τα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να έχουν ένα εργαλείο υπολογισμού της σχέσης κόστους αποτελεσματικότητας. Εμείς δεν ζητάμε να χρησιμοποιείται αυτό για τα αεροπλάνα που χρησιμοποιούνται λιγότερο, αλλά είναι, να, είναι ένα μέσο που περιφερειακά το κάθε, η κάθε χώρα να μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το δεύτερο θέμα το οποίο μας απασχολεί πολύ είναι το θέμα του ελέγχου που θα κάνει η Επιτροπή. Εμείς σεβόμαστε απόλυτα στη ρύθμιση αυτή την λήψη αποφάσεων σε περιφερειακό επίπεδο και τοπικό. Εμείς με τίποτα δεν θέλουμε να παίρνουμε τις αποφάσεις με τον ένα με τον άλλο τρόπο, εφόσον σε τοπικό επίπεδο οι αποφάσεις είναι ορθές για να αντιμετωπιστεί η χορύπηση. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο ρόλο να παίξουμε. Εμείς εδώ λέμε απλώς διαδικασίες. Προτείνουμε δηλαδή μέτρα στη ρύθμιση αυτή για να αυξήσουμε την διαφάνεια στις ρυθμίσεις που υιοθετούν οι χώρες μέλη και εφαρμόζουν. Εμείς λέμε ότι θα παρεμβαίνουμε μόνο στην περίπτωση που οι διαδικασίες αυτές δεν τηρούνται, που δεν υπάρχει κατάλληλη διαβούλευση, που δεν έχει δοθεί ο χρόνος στα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως προβλέπετε. Τη διαδικασία δηλαδή θα ελέγχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τις αποφάσεις. Ένα τελευταίο σχόλιο, επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, πολύ σύντομα για τις κατεξοδότηση πράξεις. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Πρέπει να ενημερώνουμε τις ε, διατάξεις, όπως ε, γίνεται και άλλες, ε, σε άλλες περιπτώσεις, αλλά πρέπει να μπορούμε γρήγορα να αποφασίζουμε. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και λυπάμαι που τον ξεπέρασα. Ευχαριστούμε. Όχι, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους κοιόδες εισηγητές για τα σχόλια. Θέλω να σας πω ότι και εγώ πήρα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που πήραν εκεί οι υπόλοιποι και από περιφερειακά αεροδρόμια και από εθνικές αρχές κλπ. Αλλά κυρίως από όλους τους συλλόγους εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ακόμα και μικρές ομάδες που πηρεάζονται από την κατάσταση αυτή. Γι' αυτό και προσπάθησα να παρουσιάσω μία γνωμοδότηση στην οποία να λαμβάνω υπόψη όλες τις πληροφορίες που έχω πάρει. Συμφωνώ με διάφορα σχόλια που ακούσαμε εδώ. Η ουσία της έκθεσης, και εδώ συμφωνώ με τους συναδέρφους, είναι ένα πράγμα. Η γνωμοδότηση είναι άλλο πράγμα. Οι δικές μας οι προτεραιότητες ποιες είναι, περιβάλλον και υγεία. Οι άλλες που μπορεί να είναι πιο ρεαλιστικέ στο θέμα της απόδοσης κλπ. Αυτά άλλε επιτροπές, η Επιτροπή Μεταφορών για παράδειγμα τα ασχολείται. Άρα εμείς εξετάζουμε εδώ πράγματα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των μεταφορών, αλλά έχουν να κάνουν με τι δικές μας αρμοδιότητε, που είναι η υγεία. Τα πάνε και η κυρία Κλά, η κυρία Γιανακοδάκη και άλλοι. Όλοι αναφερθήκαν στην υγεία. Πράγματι είναι υποχρέωσή μα να ε, θέτουμε προδιαγραφές για να προστατεύουμε την υγεία. Ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε. Το λίγο που μπορούμε να μετρήσουμε να το μετράμε. Λίγα πράγματα πιστεύω μας μένουν να συζητήσουμε. Το θέμα της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης, αυτό που είπε η κυρία Κλάς, κάποιες τροπολογίες μου το συμπεριλαμβάνουν αυτό το θέμα της αποτελεσματικότητας, δηλαδή. Συμφωνώ και με τις περισσότερες από τις τροπολογίες ε, Σαντών και για να Γιανακουδάκη. Νομίζω ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να ετοιμάσουμε μια καλή έκθεση. Λίγα μένουν να συζητήσουμε. Σας είπα ότι δεν θα κάνω εγώ κάσους μπέλη το αν θα είναι κανονισμός ή οδηγία. Οπότε να εκφράσω την ικανοποίησή μου που είμαστε στο σωστό δρόμο, Εμεί θα δώσουμε τη δικιά μας γνωμοδότηση και εκείνοι θα κάνουν ό,τι θεωρούν ότι πρέπει να κάνουν βάσει των δικών τους των αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Στον εισηγητή. Στάσαμε στο τέλος τη συζήτηση αυτή. Θα ψηφίσουμε 10 και 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή μεταφορά θα ψηφίσουν στις 6 Νοεμβρίου και σίγουρα θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Το θέμα του θορύβου είναι πολύ σημαντικό. Αφορά και την υγεία των ανθρώπων, των πολιτών. Το συζήτησα με τους ε, συντονιστές. Θα πρέπει να εγγύψουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη νομοθεσία. Υπάρχουν οριακέ τιμέ. Ε, πρέπει να μελετήσουμε και, την, και περαιτέρω την επίπτωση του θορύβου στην υγεία. Πρέπει να εξαντλήσουμε όλο το ερευνητικό υλικό που έχουμε στη διάθεσή μας για να μας βοηθήσει να νομοθετήσουμε. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στη συζήτηση και ξανααρχίζουμε τη συνεδρίασή μας την απογευματινή στις 3 η ώρα το απόγευμα. Ελπίζω να είσαστε πολύ άριθμοι για να συζητήσουμε το σημείο 24 της ημερησίας διάταξης όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις με την διευθύντρια, εκτελεστική διευθύντρια της ΕΦΣΑ και εν συνεχεία με την εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ε, το 26 δεν θα το συζητήσουμε, θα συζητήσουμε, θα κάνουμε μόνο τα δύο σημεία τη μέση διάταξη το 24 και 25 σήμερα το απόγευμα. Καλό διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε στις 3 η ώρα το απόγευμα.